have a list that has been sent by the political groups. Your name is not on the list, no. No, sorry. On attache number. Il y a eu un message des, des non mais c'est toujours bien. Oui. C'est un, un message qui est clair de quelqu'un. Ok. Ok. Ah oui, oui, ça va, ça va. Please, can I ask the press to let us start our meeting? Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί, λέει ο Πρόεδρος. Και επομένως, με χαρά καλωσορίζουμε σήμερα τον Μάριο Ντράγκη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για αυτό τον δεύτερο νομισματικό διάλογο του τρέχοντος έτους. Ο πρόεδρος Ντράκη θα παρουσιάσει τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τις ε, νομισματικές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερος ε, στο πρόγραμμα EPP. Ε, e, e Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει βασιζόμενο σε μία βάση ποσοτικής χαλάρωσης και επομένως έχει σαν στόχο τη δημιουργία πιο ευνοϊκών προϋποθέσεων για τον δανεισμό. Ε, το Σεπτέμβριο του 2016 ε, οπωσδήποτε θα συνεχιστεί μέχρι τότε το πρόγραμμα αυτό, το EAPP και εν πάση περιπτώσει μέχρι ότου επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τον πληθωρισμό. Ε, επίσης, ο πρόεδρος Ντράγκη εκτιμούμε ότι θα πρέπει να απαντήσει τις ε, τις ε, εξηγήσει του όσον αφορά την, ε, τον, την ομιλία της 18ης Μαΐου όσον αφορά νομισματικά ζητήματα ενός μέλους της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης καλωσορίζουμε και την επισκόπηση των επιχειρησιακών λειτουργιών όσον αφορά τα διαδικαστικά λάθη τα οποία οδήγησαν σε καθυστέρηση της ομιλίας αυτής και τώρα περιμένουμε περιμένουμε και τα νέα μέτρα και τα νέα ε, στάδια τα οποία θα καλύψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης και εξίσου σημαντικό, ο πρόεδρος Ντράγκη οπωσδήποτε θα κάνει μια αξιολόγηση όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως ε, και των ευρωπαϊκών θεσμών που έχει φτάσει σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο σήμερα. Ε, θα πρέπει ε, φαντάζομαι να μας μιλήσει και για την αρνητική έκβαση των χθεσινών συζητήσεων ε, και, την, και να καταλήξει σε μια έκκληση προς όλες τις πλευρές να ξαναρχίσουν τη συζήτηση έτσι ώστε να υπάρχει επικοδομητική προσέγγιση προς όλες τις κατευθύνσεις και να μην ακούν οι διάφορες πλευρές τις αρνητικές εκτιμήσεις διαφόρων σχολιαστών. Πιστεύουμε ότι ότι ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει και επομένως μπορεί να δώσει ε, και κάποιες ε, νέες ε, αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με υπευθυνότητα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να διατηρηθεί η ακαιρεότητα του ευρώ. Θα πρέπει όλες οι χώρες και πρωτίστως βεβαίως η Ελλάδα να δείξει και πολιτική βούληση αλλά και δέσμευση. Ε, αυτά που θα συμβούν τις επόμενες ημέρες είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους και οπωσδήποτε θέλουμε να υπάρξει ενδυνάμωση της διακυβέρνησης γιατί μονάχα μέσα από ισχυρούς θεσμούς θα μπορέσουμε ε, να λειτουργήσουμε σωστά και υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού ε, συμφέροντος. Θα ακούσουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις απόψεις του Προέδρου Ντράγκη. Πριν το λόγο στον Πρόεδρο πρόεδρο Μάριο Ντράγκη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε πρώτα μία εισαγωγική ε, παρουσίαση από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά ερωτήσεις απαντήσεις σε 5 λεπτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη καθαρχήν για την καθυστέρηση στην έλευσή μου. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που μπορώ να είμαι και πάλι ενώπιον της Επιτροπής σας για την τακτική μου συνάντηση και ακρόαση μαζί σας. Θέλω να σας παρουσιάσω την αξιολόγηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας των τωρινών οικονομικών και νομισματικών συνθηκών στη ζώνη του ευρώ. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσω το θέμα το οποίο επελέγει για την ανταλλαγή απόψεων για τα παράπλευρα αποτελέσματα του προγράμματος αγοράς αξιογράφων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα έλθω μετά και στο θέμα της τωρινή κατάστασης με την Ελλάδα η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγησή μας ότι προχωρά η οικονομική ανάκαμψη με ένα ομαλό ρυθμό, χαμηλό αλλά ομαλό ρυθμό. Η ανάπτυξη έχει υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση τα τελευταία τρίμηνα, αλλά βλέπουμε τώρα ενθαρρυντικά σημεία ότι και οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται, κάτι το οποίο υπογραμμίζει την προσδοκία μας ότι θα γίνει πιο ευρεία η οικονομική ανάκαμψη. Ιδίω θα υποστηριχθεί αυτή η πορεία από τα μέτρα μας νομισματικής πολιτικής τα οποία αρχίζουν να περνάνε στην πραγματική οικονομία. Και βοηθάει και η σχετικά χαμηλή τιμή του πετρελαίου και η βελτίωση στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά επίσης φαίνονται και στις προβλέψεις του για τη ζώνη του ευρώ. Προβλέπουμε αύξηση 1,5 μέχρι 1,9 το 2016 και να φτάσουμε σε αύξηση 2% το 2017. Μετά από πρώτους, με τους πρώτους μήνες που είχαμε αρνητικό ή μηδενικό ρυθμό πληθωρισμού, ο πληθωρισμός έχει προχωρήσει σε μικρά βήματα, είναι αυτή τη στιγμή σε 0,3% σε ετήσιο επίπεδο καθώς οι αντικές συνεισφορές των ενεργειακών τιμών πάβουν να έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει χαμηλός τους επόμενους μήνες και στη συνέχεια σε βήματα θα αυξηθεί προς το τέλος του χρόνου. Στη συνέχεια ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς επίπεδα που είναι κοντά αλλά χαμηλότερα από το 2%. Οι προβλέψεις για το ευρωσύστημα του Ιουνίου λένε ότι ο πληθωρισμός από 0,3% το 2015 θα φτάσει στο 1,5% το 2016 και 1,8% το 2017. Το τελευταίο τρίμηνο, η δυναμική των νομισματικών μεγεθών και, των, και της πίστοσης έχει βελτιωθεί. Έχουμε φτάσει σε ένα 5,3% σε νομισματική βάση και αυτό οφείλεται και στην αγορά ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα. 0,8% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα και δείχνει ότι γίνεται μεγαλύτερη σταθεροποίηση στον τομέα αυτό. Η ανάπτυξη παραμένει περιορισμένη μετά από μια φάση συρρήκνωση της ε, πιστοδοσίας και έχουμε τώρα δάνεια προς τις νέες επιχειρήσεις, τα οποία όμως είναι ακόμα ασθενικά. Γενικά παραμένουμε επιφυλακτικά ε, πεπισμένοι σε, και έχουμε την εμπιστοσύνη ότι οι οικονομικές συγκυρίες θα μπορέσουν να επιτρέψουν μια βαθμία ανάκαμψη τη, και αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωπαϊκή, στη ζώνη του ευρώ με ρυθμούς πληθωρισμού κοντά σε αλλά κάτω από το 2%. Αυτό βασίζεται στην πλήρη χρήση όλων των εργαλείων μας νομισματικής πολιτικής. Θα πρέπει να διατηρήσουμε μια σταθερή πορεία σε νομισματικό επίπεδο και να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα μέτρα και εδώ περιλαμβάνεται και το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Είναι σαφής πρόθεσή μας να αγοράσουμε ε, αξιόγραφα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα 60 ε, εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι το τέλος του, Σεπτεμβρίου του 2016 και εν πάση περιπτώσει μέχρι ότου διακριβώσουμε μια σταθερή προσαρμογή στο, στο ρυθμό πληθωρισμού που να συνάδει με το στόχο μας να επιτύχουμε ένα πληθωρισμό κάτω από το 2% αλλά πολύ κοντά στο 2% σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Τις τελευταίες εβδομάδες οι χρηματαγορές έχουν καταδείξει μια αλλαγή τάσεων σε ό,τι αφορά τις τιμές και μια αύξηση της ε, διακύμανσης με ε, σημαντικό ε, χαρακτήρα. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, η αύξηση της μεταβλητότητας, της volatility, είναι κάτι το οποίο πάντα εμφανίζεται μετά από την έναρξη ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, όταν μειώνονται οι τιμές σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Η διαδικασία ανακάλυψης τιμών είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και οι κεντρικές τράπεζες βοηθούν αυτό το φαινόμενο με την επέμβασή τους σε αξιόγραφα μεγάλης διάρκειας και βοηθούν τον τομέα των επενδυτών να κατανοήσει ποιες είναι οι πιθανές τάσεις. Επίσης, οι χρηματαγορές μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, λόγω της προσαρμογής η οποία εισήχθη ακόμα και πριν από το διευρυμένο πρόγραμμα μας αγοράς αξιογράφων που ξεκίνησε το Μάρτιο του ελεστώτος έτους, η, τα επιτόκια, τα διατραπεζικά επιτόκια που είναι κύριος δείκτης για τις οικονομικές συνδίκες στην αγορά της Ευρώπης κινούνται ακόμα προς τα κάτω. Μετά από την διακήρυξη του διευρυμένου αυτού προγράμματος αγοράς αξιογράφων, ο σύνθετος, το σύνθετο επιτόκιο για τις ε, δανειοδοτήσεις μη χρηματοπιστωτικών εταιριών μειώθηκε στο 2,3% τον Απρίλιο, δηλαδή μειώθηκε κατά 13 εκατοστία στοιχεία που είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιούνιο του 2013. Επίσης, τα δάνεια προς ε, νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 25 σε εκατοστία στοιχεία στο 2,5 τον Απρίλιο έναντι 2,8 που ήταν τον Ιούνιο του 2014. Επιπλέον, τα περισσότερα, οι περισσότεροι δείκτες διασποράς δείχνουν σημαντική μείωση σε ό,τι αφορά τις μη χρηματοπιστούν χαρατήρα εταιρείε. Όσοι έχουν τώρα τα επιτόκια τροποποιούνται οι συμφωνίες δανειοδοτικού χαρακτήρα, αντικαθιστούν νέες πιο ευνοϊκές συμφωνίες στις προηγούμενες και η προσαρμογή σε χρηματοοικονομικό επίπεδο πλησιάζει περισσότερους επενδυτές και καταναλωτές. Αυτή η σταδμία, σταδιακή διαδικασία δεν έχει περατωθεί ακόμα, συνεχίζεται. Τούτου όμως λεχθέντος, στη διαδικασία της προσαρμογής των τιμών, η μορφή των επιτοκίων σε χρονικό επίπεδο έχει υποστεί μεγάλη πίεση. Η πολιτική η οποία θα έπρεπε να προκύπτει από την εικόνα της αγοράς έχει οδηγήσει στην καμπύλη απόδοσης να γίνεται πιο απότομη. Η πλευρά της καμπύλης αυτής που αφορά τις ε, βραχυπρόθεσμες ε, προσδοκίες λόγω της αύξησης της ρευστότητας έχει παραμείνει στο ίδιο επίπεδο σε επίπεδα τα οποία ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ε, καθοδήγηση που δίδει η Κεντρική Τράπεζα. Παρακολουθούμε προσεκτικά τις ε, συνθήκες για να δούμε να, μήπως υπάρξει ανάγκη να αντιδράσουμε σε μια υπερβολική ε, σε ό,τι αφορά την παροχή ρευστότητας από τη δική μας πλευρά. Τώρα ερχόμαστε στα παράπλευρα αποτελέσματα του προγράμματος αγοράς αξιογράφων υπάρχουν κίνδυνοι που ελοχεύουν σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλω να εστιάσω περισσότερο στους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην περιοχή του ευρώ και τα αποτελέσματα για την κατανομή εισοδήματος στην ίδια ζώνη. Εμείς παρακολουθούμε τον κίνδυνο για τον ισολογισμό της ζώνης του ευρώ που επηρεάζεται από τις αγορές αξιογράφων ώστε να μην εμποδίσουμε την ικανότητά μα να κρατήσουμε τη σταθερότητα των τιμών, που είναι και η εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμεί θέλουμε να διαχειριστούμε του κινδύνου ε, σε πιστοτικό επίπεδο με το να έχουμε αξιόγραφα επαρκού ποιότητος, με το να έχουμε περιορισμού σε σχέση με τι αγορέ αυτέ, που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τι αγορέ αυτέ, και με το να, να έχουμε την πρέπουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογή των αξιογράφων σε ό,τι αφορά το PSPP, το, δηλαδή τα κρατικά αξιόγραφα, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα εφαρμοστεί από, τα, από τις κεντρικές τρέπεζες των κρατών μελών δεν θα οδηγήσει σε διαμερασμό κειμένου κινδύνου με το σύστημα του ευρώ. Αυτό δεν περιορίζει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού και την ενιαία κατεύθυνση της νομισματικής μας πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη ε, εικόνα όλης αυτής της διαδικασίας και λαμβάνουμε υπόψη την ενιαία ε, δομική ε, αντιμετώπιση μιας ενιαίας πολιτικής η οποία μπορεί να συνάδει και να συμβαδίζει με τις 19 εθνικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κινδύνους σε επίπεδο χρηματοπιστικής σταθερότητας, θεωρούμε ότι αυτή η κίνδυνη είναι προς το παρόν περιορισμένη. Αν δούμε ιδιαίτερα την στεγαστική αγορά στην ζώνη του ευρώ, δεν βλέπουμε στοιχεία του να υπάρχει διόγκωση των τιμών. Υπάρχουν σημαντικοί δείκτες για την αύξηση των ε, ε ανισομεριών που κυρίως απεικονίζονται στις τιμές των ακινήτων και στις τιμές των αξιογράφων. Βλέπουμε παραγωγός χάρη ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της τιμής στο στεγαστικό τομέα είναι 0,5% στο τελευταίο τρίμηνο του 2014. Για τις ε, στεγαστικές υποθήκες, ο ρυθμός αντίστοιχος είναι 0,1% τον Απρίλιο του 2014. Παρακολουθούμε λοιπόν όσες αυτές τις εξελίξεις και γι' αυτό η μακροπολιτική μας πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι παραμένει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τέλος, οι μεγάλες κλίμακος αγορές αξιογράφων όπως και οπουδήποτε άλλο μέτρο νομισματικής πολιτικής έχουν και επιπτώσεις στη διανομή του πλούτου. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ο τωρινός συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων και της ε, κατεύθυνση που δίνει η Κεντρική Τραπέζα και, τα, και της αγοράς ομολόγων θα οδηγήσει σε αύξηση των ε, τιμών των ε, ε, στοιχείων ενεργητικού και θα αυξήσει τον πλούτο αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι αυτών των στοιχείων ενεργητικού. Αλλά αυτή η αύξηση ε, είναι και ένας τρόπος μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και φυσικά κινητοποιείται κάθε φορά που μια κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τα εργαλεία της νομισματικής πολιτικής της. Είτε είναι συμβατικά ή μη συμβατικά τα εργαλεία αυτά νομισματικής πολιτικής. Οι αλλαγέ των επιτοκίων πάντα αλλάζουν την ελκυστικότητα της αποταμίευσης εναντί της κατανάλωσης και μπορούν να επηρεάσουν και το βάρος του χρέους των δανειστών. Ως έχουν λοιπόν τα πράγματα, εμείς έχουμε σαν στόχο να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση σε επενδύσεις και σε κατανάλωση στην οικονομία που θα οδηγήσει και σε υψηλότερο πληθωρισμό. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουν τα επιτόκια να επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα τα οποία να συνάδουν με μια βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα των τιμών. Με την μείωση του κυκλικού στοιχείου του υπερκυκλικού στοιχείου της απασχόλησης μπορούμε έτσι να μειώσουμε και μια σημαντική πηγή ανισότητας σε επίπεδο εισοδήματος. Η νομισματική μας πολιτική οδηγεί λοιπόν σε αυτή τη μείωση της ανισότητας, ιδίως μεταξύ των νέων και αυτών που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Σε τελική ανάλυση όλοι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ θα αποκομίσουν ωφέλη από ένα περιβάλλον σταθερών τιμών, μακροοικονομικής σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Να πω και κάτι τώρα για την τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσοι έχουν τα πράγματα για οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ζώνης του ευρώ μάλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει να εκτελέσει την εντολή της ως Κεντρική Τράπεζα και έναντι της Ελλάδος. Επιπλέον, οι κανονισμοί του ενιαίου μηχανισμού τραπεζικής εποπτείας που ενεκρίθησαν κάνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επόπτη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και άμεσα και έμεσα μέσω της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας. Μέσα στο δίπτυχο το TUPAC, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει από την Κομισιόν να είναι σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν γίνονται οι διαπραγματεύσει για την αιρεσιμότητα η οποία συνοδεύει το πρόγραμμα προσαρμογή και όταν παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματο αυτού. Όταν πρόκειται λοιπόν για την νομισματική πολιτική και τι εποπτικέ δραστηριότητε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσει με απόλυτη ανεξαρτησία και ακολουθώντα το νομικό πλαίσιο που τη διέπει. Αυτή η προσέγγιση βάση κανόνων είναι αυτό το οποίο απαιτείται από τη δική μα πλευρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμεί έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα και αυτή θα είναι η πορεία μα και στο μέλλον. Μέσα στο πλαίσιο αυτό το σύστημα το η ζώνη του ευρώ έχει δώσει υποστήριξη για να συνεχίσει να δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία. Η ρευστότητα της κεντρικής τράπεζας, η οποία έχει δοθεί στις ελληνικές τράπεζες, φτάνει περίπου το 118 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου διπλάσιο το ποσό το οποίο είχε δοθεί μέχρι το 2014. Η τωρινή υποστήριξη σε επίπεδο ρευστότητα είναι 66% περίπου του ΑΕΠ της Ελλάδος. Είναι το υψηλότερο επίπεδο ως μερίδιο του ΑΕΠ που υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα της ζώνης του ευρώ. Την προηγούμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να μην θέσει αντιρρήσεις σε περαιτέρω αύξηση στην οροφή του ELA, της πρόσθετης ε, ενίσχυσης ρευστότητος για να φτάσουν τα 83 δισεκατομμύρια η έκτακτη βοήθεια. Θα συνεχίσει λοιπόν αυτή η βοήθεια ρευστότητα, όσο είναι φερέγγιε οι ελληνικέ τράπεζε και έχουν επαρκή στοιχεία εγγύησεων. Εάν όμω η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πρόσβαση στην αγορά, αυτή η ρευστότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2.3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί λοιπόν με τις ανάγκες της εποπτείας εξηγούν γιατί υπάρχει ανώτατο όριο για τα ελληνικά ομόλογα, τα, οποία, τα κρατικά ομόλογα τα οποία μπορεί να έχει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Για να εξεταστεί αυτή η οροφή για τα κρατικά ομόλογα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική για επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων και την μελλοντική του εφαρμογή, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουν να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια από την <clears throat> από τους ευρωπαϊκούς φορείς. Αυτό φυσικά θα βελτιώσει ιδιαίτερα και την προσδοκή, προσδοκία μελλοντικής πρόσφασης της αγοράς από την ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η απόφαση για το αν θα περατωθεί η εξέταση του τωρινού προγράμματος και, θα, και αν θα απελευθερωθούν περαιτέρω κονδύλια προς την Ελλάδα, αυτό βρίσκεται στα χέρια της Ευρωομάδος. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στη ζώνη του ευρώ να αποφασίσουν. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί από εκλεγμένους λήπτες αποφάσεων και όχι από τους κεντρικούς τραπεζίτες. Ενδιαμέσως στο ενδιάμεσο διάστημα θα συνεχίσουμε να δίνουμε συμβουλές για το πρόγραμμα προσαρμογής και μέσα στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να έχουμε μια στεναρή και πλήρη συμφωνία με την Ελλάδα και χρειάζεται αυτό να γίνει πραγματικότητα πολύ σύντομα. Και ισχυρή και πλήρη σημαίνει μια συμφωνία η οποία θα οδηγήσει σε ανάκαμψη, η οποία έχει κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά είναι και δημοσιονομικά εφικτή και βιώσιμη. Εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα, αντιμετωπίζει τις περαιτέρω πηγές ε, χρηματοοικονομικής ασταθείας και δημοσιονομικής αστάθειας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να εξασφαλίσει μια τέτοια επιτυχή έκθεση. Μια τέτοια ισχυρή και αξιόπιστη συμφωνία με την Ελλάδα χρειάζεται όχι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδος, αλλά και προς το συμφέρον όλης της ζώνης του ευρώ όλοι οι εμπλακόμενοι θα πρέπει να κάνουν περαιτέρω προσπάθειες για να φτάσουμε σε μια λύση, αλλά η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ευρωπα... ελληνικής κυβέρνησης που θα πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Η κατάσταση στην Ελλάδα μας θυμίζει και πάλι ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ημιτελής όσο δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη της ζώνης του ευρώ μπορούν να είναι οικονομικά, δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά αρκετά ανθεκτικά. Για να μπορέσει να συμπληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση χρειαζόμαστε ένα ποιοτικό άλμα προς ένα ισχυρότερο ε, θεσμικό πλαίσιο, μια ισχυρότερη θεσμική αρχιτεκτονική. Όπως ξέρετε οι συνάδελφοί μου και εγώ ε, εργαζόμαστε για μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει ε, μια πρόταση οδικού χάρτη προς την κατεύθυνση αυτή. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της εκπόνησης αυτής της έκθεσης και ελπίζω ότι θα κατανοήσετε ότι και από σεβασμό για τους συναδέλφους μου, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα από αυτά που έχω ήδη πει στο παρελθόν. Ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο στεναρό θεσμικό πλαίσιο για να κάνουμε αυτή την ποιοτικ... αυτό το ποιοτικό άλμα που ανέφερα προηγουμένως και προσβλέπω τώρα στα ερωτήματά σας. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Ντράγκη για τα σοφά και σημαντικά σας λόγια. Ευελπιστώ ότι όλοι τα άκουσαν με τη δέουσα προσοχή και τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρώτο μιλητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας και κυρίως για την δουλειά που έχετε κάνει ιδιαίτερα στους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η παρουσίαση αφήνει πολλά ερωτηματικά και θα ήθελα να περιοριστώ σήμερα σε δύο ερωτήματα για να μπορέσετε να έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Καταρχάς, αναφερθήκατε στα, στις πιστώσεις έκθεσης ρευστότητας, 118 δις ευρώ συνολικά, χωρίς ανώτατο όριο ως τώρα. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσον μπορείτε να επεξηγήσετε πιο λεπτομερώς υπό ποιους όρους έχουν δοθεί αυτά τις επιστώσεις τους τελευταίους ε, μήνες και εβδομάδες, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Κατά δεύτερον, δεύτερη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας, ΑΙΟΠΑ, τονίζει όλο και πιο πολύ ότι τα ακραία επιτόκια επιβαρύνουν και τις ασφάλειες αλλά και όλους τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Θα ήθελα να ακούσω κατά πόσο η δική σας στρατηγική σημαίνει ότι προωθούνται τα βραχυπρόθεσμα μέτρα εις βάρος των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων μέτρων. Thank um, Σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση για το ELA, για την εκτρευστότητα. Αυτό χορηγείται στις τράπεζες που είναι φερέγγιες, αυτή η έκδοτη και σε τράπεζε που έχουν τη να παρέχουν επαρκή εχέγγυα. Η εκτίμηση του υποπτή είναι ότι στη φάση αυτή οι ελληνικέ τράπεζε είναι φερεγγίε. Οι μεγάλε ελληνικέ τράπεζε. Και ω εκ τούτου, οι εγγυήσει που παρέχουν επαρκούν. Ασφαλώς. Η κατάσταση είναι εν εξελίξη. Και άρα, όπως κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στενά. Για να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι όροι για την αξιολόγηση των εχηγείων εξακολουθούν να είναι οι ίδιες και γενικότερα να αξιολογούμε την υγεία των τραπεζών. Δεν υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο όριο για το ELA, για αυτή την αρρωγή ρευστότητα. Αυτό εξαρτάται από τη φερεγγιότητα τη τράπεζα και από τα εχέγγυα που παρέχονται. Για το δεύτερο ερώτημα. Ανταλαμβανόμαστε ότι η ΟΠΑ έθεσε το θέμα αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Έχουμε μία εντολή. Η εντολή είναι να υπάρξει μία εποπτική πολιτική που θα ακολουθεί το στόχο της σταθερότητας των τιμών με συντελεστή πληθωρισμού κάτω από 2%. Αυτή είναι η εντολή μας. Αν τώρα υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα με τις ασφαλιστικές, με τους μακροπρόθεσμους επενδυτές χαμηλού επιτοκίου ή γενικά αν υπάρχει τέτοιος χρηματοοικονομικός κίνδυνος, θα αξιολογήσουμε τον κίνδυνο, θα παρακολουθήσουμε τα πράγματα και όπως σας είπα πριν από λίγο δεν βλέπουμε να διακρίνεται τέτοιος κίνδυνος ιδιαίτερος. Αλλά Μπορούμε ασφαλώς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την νομισματική πολιτική. Θα ήταν λάθος να κάνουμε κάτι που ξέρουμε ότι αποτελεί λαθασμένη νομισματική πολιτική μόνο και μόνο για τις ασφαλιστικές. Είναι ασφαλώς περίπλοκα τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι το εξής. Οι ασφαλιστικές δεν είναι όλες οι ίδιες. Τι σημαίνει αυτό η αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ ε, των ε, αξιογράφων και των ευθυνών είναι πολύ πιο υψηλός για κάποιες ε, ασφαλιστικές από κάποιες χώρες και πολύ πιο χαμηλός για κάποιες άλλες ασφαλιστικές από άλλες χώρες. Και αυτό εξαρτάται, δηλαδή ο μακροπρόθεσμος αντικτύπος των επιτοκίων εξαρτάται και από το επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο ισχύει. Είναι σαφές ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που δίνουν σταθερά ε, επιδόματα έχουν πιο μεγάλη έκθεση με μακροπρόθεσμα επιτόκια και εξαρτώνται πολύ πιο πολύ από τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Η ΟΠΑ δεν εκτιμάει ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος άμεσα σε ορίζοντα 6 έως 10 έτη. Είναι ασφαλώς κάτι που μας απασχολεί, αλλά δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Τέλος, οι ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ και κάποιο καιρό έχουν αντιδράσει στην κατάσταση αυτή αναζητώντας επενδύσεις σε αξιόγραφα τα οποία διαφέρουν από αυτά στα οποία επένδυνε ως τώρα. Είναι μια αργή διαδικασία η οποία θα καθοδηγήσει τις επενδύσεις σε τομείς αναγκαστικά πιο επικίνδυνους, ίσως και με λιγότερη ρευστότητα, και στη φάση αυτή πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Προσπαθούμε δηλαδή να αυξήσουμε την απόδοση στις επενδύσεις των ασφαλιστικών. Έχει έρθει όμως η στιγμή να σκεφτούμε κατά πόσον αυτή η διαδικασία διαφοροποίησης των επενδύσεων έχει βοηθήσει, έχει αποφέρει καρπούς βάσει του υφιστάμενου κανονισμού ή κατά πόσον έχει αποτραπεί μάλλον, εμποδιστεί από τους υφιστάμενους κανονισμούς. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό. Ευχαριστώ. Και η Επιτροπή αυτή, λέει ο Πρόεδρος, έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Και αυτό αναγνωρίζεται και στον οργανισμό ΕΦΣΥ. Η Ελίζα Φερέιρα είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετίζω και πάλι ανάμεσά μας. Θα ήθελα να παραθέσω καταρχήν αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το πρόβλημα της Ελλάδος θα πρέπει να επιληθεί σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αναφερθεί ως ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος αυτού. Δεν αναφερθήκατε στα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να απελευθερωθούν επί τη βάση αυτής της συμφωνίας. Δεύτερον, είπατε ότι αν υπήρχε στάση πληρωμών από την πλευρά της Ελλάδος, δεν θα υπήρχε καμία επιμόλυνση μέσα εισαγωγικά της ζώνης του ευρώ. Έχετε την απόλυτη βεβαιότητα όμως ότι υπάρχει η απόλυτη προστασία από κίνδυνους επιμόλυνσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εξασφαλισμένο κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ιστορικά, αν δούμε τα πράγματα, αν υπάρξει μια στάση πληρωμών, η ευρωπαϊκή ζώνη του, η ζώνη του ευρώ ουσιαστικά διασπάται. Και από ό,τι έχω υπολογίσει θα υπάρξει μια απώλεια που θα φτάσει το 0,02% του ΑΕΠ της σύνολης ευρωπαϊκής ζώνης. Τη στιγμή λοιπόν που εσείς αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν ήδη ελλείψεις στην ευρωπαϊκή νομισματική αρχιτεκτονική, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύετε αυτή τη δήλωσή σας που είναι τόσο σημαντική ότι το ευρώ θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να διατηρηθεί η ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ, του ευρώ με κάθε τίμημα στη συγκεκριμένη περίπτωση της κρίσης Ελλάδος. Ευχαριστώ λέει κύριε Στράγγι. Επιτρέψτε μου πρώτα να πω κάτι το οποίο ε, ίσως ε, χρειαστεί να επαναλάβω πολλές φορές σήμερα και το λέω, το πολύ συχνά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι πολιτικό θεσμικό όργανο. Αυτό σημαίνει ότι ε, δρά, ενεργεί σύμφωνα με υφιστάμενους κανόνες. Δεν δημιουργούμε νέους κανόνες εξ νόβο λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα συγκυρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ρόλος μας είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που ε, έχουν τα κράτη της Ευρωζώνης. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου από την κυρία Φερέιρο. Ναι, εντάξει, απαντάω ο κύριος Δράκη, εγώ απαντώ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είπατε ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιμόλυνσης. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους οικοτολογίες, ε, ε, ούτε να αναφερθώ σε μελλοντικές ε, υποθετικές εκβάσεις της κατάστασης. Σίγουρα δεν θέλουμε να μπούμε σε αχαρτογράφητα, αχαρτογράφητα ύδατα, γιατί εμείς λέμε και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε όλα τα εργαλεία έτσι ώστε να μας επιτραπεί να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα την κατάσταση, όπως άλλωστε έχουμε κάνει μέχρι τώρα και σε άλλες ε, περιστάσεις, ενδεχομένως όχι τόσο ε, δραματικές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποιε ε, θα είναι οι μέσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο τούτη τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε, ούτε μπορούμε να το σχολιάσουμε υποθετικά. Είναι πάντως σαφές ότι ε, τα τεκτενόμενα καταδεικνύουν ότι είναι ημιτελής ε, η κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις οποιοδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος μεγάλου εύρους, οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, ε, κάνουμε αυτό το quantum leap, το ποιοτικό ε, άλμα και θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιες ακριβώς περιοχές θα πρέπει να λάβει χώρα αυτό το άλμα. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, το EFSF έχει κανόνες βεβαίως και δίνει συγκεκριμένε δυνατότητες ε, στα κράτη-μέλη. Ε, ο κύριος Μαριάς από το ΙΣΙΑ. E ε, Θα μιλήσω στα ελληνικά κύριε Ντράγκη, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. ορίσω στην Επιτροπή μας. Έθελα να επισημάνω ότι η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται στο 26,6% και η ανεργία των νέων χτύπησε κόκκινο, φτάνοντας το 51,7% σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την περασμένη Παρασκευή. Το 40% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το 45% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη κάτω από 650 ευρώ και το ελληνικό δημόσιο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του προς τρίτους. Κύριε Ντράγκη, σας διαβάζω το άρθρο 7 του κανονισμού 3603 του 1993 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου του 1993 το οποίο αναφέρει επιλέξει τα εξή. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες προς το δημόσιο τομέα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν θεωρείται πιστοτική διευκόλυνση κατά την έννοια του άρθρου 104 της Συνθήκης. Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας για την αποπληρωμή των δανείων του Δούνου που έλαβε το Μάιο του 2010 με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αδυναμία πληρωμής θα ήθελα να σας ρωτήσω ως πρόεδρο της ΕΚΤ ποια θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση αξιοποιώντας το άρθρο 7 του κανονισμού 3603 του 1993 ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δανειοδότηση της ελληνικής δημοκρατίας για τη μερική ή ολική εξόφληση των παραπάνω δανειακών υποχρεώσεων της έναντι του Δουνουτού, το οποίο Δουνουτού σύμφωνα με τελευταίες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις έχει τορπιλήσει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών. Να σημειώσω εν προκειμένου ότι εσεί ο ίδιο ω διοικητή έχετε δώσει την έγκρισή σα σε ανάλογε περιπτώσει που αφορούν την Ιταλία, την οποία έχω εδώ μπροστά μου, την Αυστρία δύο φορέ, την Πορτογαλία, ενώ ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας, κατόπιν άδεια του κυρίου Τρισέ, δανειοδοτήσατε την Ιταλική κυβέρνηση για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Δέλτα Νιτάφ. Έχω εδώ τις αποφάσεις. Εν ώψη του ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και τελειώνω, βάσει των συνθήκων, μεριμνά ώστε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες να τηρούν τις εκ της συνθήκης υποχρεώσεις ποια θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν 10 seconds, Mr. Chairman. Ποια θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη Εθνική Κεντρική Τράπεζα της Ευρωζώνης προχωρήσει στη δανειοδότηση της ελληνικής δημοκρατίας προκειμένου να προβεί σε μερική ή ολική εξόφληση των υποχρεώσεων της προς το Δέλτα Νιτάφ. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή δραματική, κυρίως δε αν αναφερθούμε στην ανεργία, κυρίως δε ανεργία των νέων. Όπως γνωρίζετε και απαντώ τώρα στην ερώτησή σας, ε, υπάρχει το άρθρο 123 ε, της συνθήκης ε, που λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε πιστοτική διευκόλυνση αλλά θα ήθελα να κάνω μια, ένα γενικότερο σχόλιο παρατήρηση του κ. Μαριά εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς δυστυχώς. Oh. Can I, can I, yeah, I mean, just, uh, I wouldn't agree with your δεν μπορώ να συμφωνήσω με την εξαίρεση που αναφέρατε, αλλά θα ήθελα να κάνω ακόμα ένα γενική φύσεως σχόλιο, γιατί φαίνεται ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα ε, φαίνεται σαν να είναι, ε, ε, σαν να είναι ευθύνη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν δίνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, εγώ επανειλημμένα έχω δώσει όλη την, όλο το ιστορικό των χρηματοπιστωτικών ροών προς την ε, ε, Ελλάδα. Έχουμε δει ότι πολυμερή και διμερή δάνεια, ε, καθώς επίσης και οι καθαρές μεταφορές, καθώς επίσης και άλλου είδους μεταφορές. Στα πλαίσια του μηχανισμού ε, σταθερότητας φτάνουν σε πάνω από 200 εκατομμύρια ε, ευρώ, 223 συγκεκριμένα, τα οποία είναι ε, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουμε παράσχει χρηματοδότηση και στήριξη στο, ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 118 εκατομμύρια, ε, δηλαδή 66% του ΑΕΠ της ε, Ελλάδος. Εδώ θα πρέπει να προσθεθούν και τα ε, χρήματα από τον μηχανισμό στήριξης IMF, καθώς επίσης και το κούρεμα το οποίο έλαβε χώρα στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης του χρέους και που αποτελούσε περίπου 53% του ε, ΑΕΠ ε, δεν θέλω βεβαίως να δώσω υπερβολική ε, σημασία σε αυτούς τους αριθμούς που όμως έχουν ιδιαίτερο βάρος. Θα ήθελα απλώς να δείξω ότι η δραματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι ε, για, την, ε, αυτήν την κατάσταση. Κοιτάξτε, εμείς σας λέμε ότι κάνατε κάτι αντίστοιχο στην στην περίπτωση της Ιταλίας Πρόεδρος, αγαπητέ συνάδελφε, δεν μπορείτε να διακόπτετε τον Πρόεδρο. Εγώ αναφέρθηκα ε, στον ε, κανονισμό 3603. Κύριε Μαριά, ξέρετε ότι, λέει ο Πρόεδρος, ότι, το, ότι ο κανονισμός αυτός υπόκειται σε περιορισμούς βάσει του άρθρου 123 των συνθήκων. Ναι, αλλά λέει ο κύριος Μαριάς, αυτός ο κανονισμός 3603 του 1993 έχει ήδη εφαρμοστεί. Πρόεδρος, θα πρέπει να διαβάσετε καλύτερα και σωστότερα τον κανονισμό αυτό, ο οποίος υπόκειται σε άλλους περιορισμούς. Ο κύριος Ντράγκη, είμαι απολύτως ε, έτοιμος να ε, ε, μιλήσω μαζί σας για το θέμα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς σας υπέβαλα αυτό το ερώτημα, κύριε Ντράγκη, ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρος, αυτός ο κανονισμός υπόκειται στην εφαρμογή του σε ορισμένες διατάξεις οι οποίες ρετά αναφέρονται στο άρθρο 123. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μαριάς, θα πρέπει να διαβάσετε τον, τον κανονισμό αυτό σωστά και να μην κάνετε τέτοιου είδου υποθέσει. Καλησπέρα κύριε Τράκη. No, thank you. Thank you, Mr. President, for... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και για όλα αυτά που κάνετε για μας. Παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που κάνετε για την Ευρώπη και υποστηρίζουμε τις προσπάθειές σας για να είσαστε επικοδομητικός και για να τηρήσετε και τους κανόνες, αν μου επιτρέπετε. Να τηρήσετε τους κανόνες για την δικαιοσύνη και την αξιοπιστία. Αλλά ανησυχώ. Είπατε επανελειμμένα και στο Ελσίκη και στη Φραγκφούρτη και στη ε, ημερίδα της Deutsche Bank ότι είμαστε ημιτελείς ως Οικονομική Ένωση και ότι θέλουμε μια ένα ποιοτικό άλμα. Είσαστε σίγουροι ότι οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν τι σημαίνει το ποσοτικό αυτό άλμα και μήπως κάνουν ό,τι μπορούν για να πετύχουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αν χάσουμε ένα κράτος μέλος ή αν υπάρξει στάση πληρωμών. Πολύ φοβάμαι ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση των επενδύσεων και για την ανάπτυξη θα, πάνε, θα πέσουν στο νερό. Ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένο ε, ακόμη ότι χρειαζόμαστε αυτό το ποιοτικό άλμα. Επίσης, πεπισμένο είμαι ότι η κατεύθυνση αυτού του άλματος είναι σαφής σε γενικές γραμμές. Και ως εκ τούτου είναι κατανοητό. Τούτου λεχτέντος. Θα πρέπει να σεβαστούμε τους διαφόρους ρόλους. Ποιος είναι ο ρόλος μας εδώ? Να πούμε τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα αυτό, να καταστεί πιο ανθεκτικό προκειμένου να διορθώσουμε τις αδυναμίες τους. Μία μόνο εξ αυτών είναι η Ελλάδα. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε διάφορα παραδείγματα για το πόσο ευάλωτη είναι αυτή η Ένωση. Άρα καθήκον μας στο σημείο αυτό είναι να υποδείξουμε το τι θα πρέπει να γίνει. Το καθήκον των κρατών μελών, των κυβερνήσεων τους, είναι να ηγεθούν. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το καθήκον υπό κάποια έννοια να περάσουν τις αλλαγές αυτές από το εκλογικό σώμα, να εξηγήσουν τις αλλαγές αυτές, να εξηγήσουν και το δυναμικό και τα ωφέλη σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, τα ωφέλη ενός ε, τελείου συστήματος, ολοκληρωμένου συστήματος. Θα έλεγα ότι κάποιες από τις θυσίες, ένα ποσοστό της φτώχειας, της ανεργίας που δημιουργήθηκε ως απόρρια της μεγάλης κρίσης που είχαμε το 2009 προήλθε από το γεγονός ότι αυτό το οικοδόμημα ήταν ημιτελές. Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που μου είπατε και καλησπέρα. Thank you for... Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο Μίκελ Ουτμπάν έχει το λόγο. Όπως ξέρετε πολύ καλά, και καταρχήν να σα ευχαριστήσω πρώτα για την παρουσία σας κύριε Ντράγκη. Αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, το ΑΕΠ της Ελλάδος έχει μειωθεί κατά 25% από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο. Ένας οικονομικός αντίκτυπος ο οποίος είναι χωρίς προηγούμενο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα οικονομικό πόλεμο όπου η κυριαρχικότητα και η ελευθερία του ελληνικού λαού βρίσκεται υποκίνδυνο. Βάσει της έκθεσης για τον έλεγχο του ελληνικού χρέους που έχει γίνει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα παρουσιαστεί την επόμενη Πέμπτη στην Πέμπτη, υπήρξαν σημαντικές ατασταλίες σε ό,τι αφορά την διαχείριση του ελληνικού χρέους από την προηγούμενη Τρόικα. Από το Σεπτέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει απεριόριστα αξιόγραφα κρατικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του συστήματο ε, οριστικών χρηματοοικονομικών αγορών. Αλλά δεν έχει αγοράσει κανένα ελληνικό ομόλογο. Έχετε εξαρτήσει αυτήν την αγορά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που δεν είναι δημοκρατικός φορέας και εξαρτάται από τα πολιτικά συμφέροντα των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας. Κύριε Τράγκη, μήπως με τον τρόπο αυτό παραβιάστε το άρθρο 130 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίρνει εντολές εκ των έξω. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό στην περίπτωση αυτή ένα μη δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο δίδει κατευθύνσεις και δεν επιτρέπει στην Ελλάδα την πρόσβαση στο σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης από το Μάρτιο του 2015 που συμπίπτει ως εκτύχης με την ε, ανάρρηση στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ντράγκη. Μήπως αυτό δεν αποτελεί μια διάκριση με πολιτικό χαρακτήρα που ουσιαστικά οδηγεί την Κεντρική Τράπεζα να παραβιάσει την αρχή της ουδετερότητας η οποία πρέπει να την διέπει, κύριε Ντράγκη. Μήπως χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή η Κεντρική Τράπεζα ως εργαλείο εκβιασμού στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδος και των Ευρωπαϊκών Θεσμών και της ομάδας των Βρυξελών και με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η κυριαρχικότητα του ελληνικού λαού που έχει εκφραστεί στις εκλογές 25 Ιανουαρίου. Γιατί η κρίση της ε, ε, έχει οδηγήσει σε 20% αύξηση της αυτοκτονίας. Δύο σε κάθε πέντε παιδιά στην Ελλάδα είναι κάτω από το επίπεδο της ένδυας. Πάρα πολλοί δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Κύριε Δράγη, μήπως θεωρείτε ότι όλα αυτά δεν είναι ένα πανόραμα οικονομικού πολέμου και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα οικονομικών αποφάσεων οι οποίες επιβάλλονται αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Ποια είναι η ερώτησή σας? Σας έκανα τρεις ερωτήσεις. Αν θέλετε μπορώ να τις επαναλάβω. Well, κύριος Ντράκη. Η ερώτησή σας θεωρώ είναι ότι γιατί δεν αγοράζουμε τα ελληνικά ομόλογα και γιατί δεν συμμετέχει η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση. Τρεις είναι οι λόγοι και να σας πω εν παρόδο ότι όλα αυτά ε, ε, προϋπήρχαν της ελληνικής κρίσης και η λύση ε, βαδίζει βάσει προϋφισταμένων στοιχείων. Επομένως δεν πρέπει να βρείτε στη δικιά μας δράση κάποιες πολιτικές ας πούμε διαστάσεις. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό όργανο. Εμείς είμαστε ένας θεσμός ο οποίος βασίζεται τη λειτουργία του σε κανόνες και εμείς με συνεκτικό τρόπο πάντοτε εφαρμόζουμε εφαρμόζουμε τους κανόνες αυτούς. Τώρα, εάν θέλετε να με ρωτήσετε γιατί δεν αγοράζουμε ελληνικά ομόλογα στα πλαίσια της προσωπικής χαλάρωσης, η απάντησή μου είναι η εξής δεν αγοράζουμε ομόλογα από χώρες ε, οι οποίες ε, βρίσκονται ακόμα ε, σε μη ολοκληρωμένη αξιολόγηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην περίπτωση της Κύπρου επίσης το είχαμε εφαρμόσει αυτό. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που το κάνουμε. Δεύτερον, δεν αγοράζουμε ομόλογα τα οποία βρίσκονται κάτω από ένα ποσοστό το οποίο των οποίων η ποιότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ε, μονάχα εάν ε, υπήρχε ένα waiver σε αυτά τα ομόλογα ε, τότε θα μπορούσαμε να τα είχαμε αγοράσει. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη την αγορά της Ελλάδος δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι η πρώτη φορά Τώρα, ε, όσον αφορά αυτό που είπατε στο τέλος, δεν αγοράζουμε περισσότερο από 23% ε, κρατικών ομολόγων ε, για τις οποίες έχουμε ήδη ευρωομόλογα. Δηλαδή, μπορούμε μονάχα να αγοράσουμε, και το έχουμε κάνει για την Ελλάδα, ορισμένο ποσοστό των ομολόγων. Αυτές είναι, επομένως, οι τρεις προϋποθέσεις τις οποίες σας ανέφερα, δηλαδή να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ε, να μην υπάρχει το waiver και ενδεχομένως να ε, μην ε, αλλάξει η ποιότητα ας πούμε των ομολόγων. Εάν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις δεν συντρέχουν, δεν είναι δυνατόν να αγοράσουμε ελληνικά ομόλογα. Μονάχα εάν ολοκληρωθούν αυτές οι τρεις διαδικασίες και αν υπάρξει και η πολιτική απόφαση, εμείς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την στάση δεν μπορώ εγώ να αξιολογήσω τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο ε, όταν θα στεφθούν από επιτυχία αυτές οι διαπραγματεύσεις, ε, τότε αυτές οι προϋποθέσεις θα έχουν πληρωθεί και επομένως θα μπορέσουμε... Άρα αναγνωρίζετε τον εκβιασμό από τους πράσινες, η ομιλητρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα σας ρωτήσω για την Ελλάδα, θα σας ανακουφίσει αυτό. Θα σας ρωτήσω για τις παράπλευρες απώλειες του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Τρία χρόνια, λοιπόν, μετά την έναρξη της προσωπικής χαλάρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Αγγλίας υπολόγισε ότι μειώθηκε η αξία των αξιογράφων κατά 26% λόγω της πολιτικής. Και αυτό σημαίνει ότι 40% των κερδών πήγε στα πιο πλούσια νοικοκυριά. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά η ποσοτική χαλάρωση αύξησε τις, ε, τα χάσματα για να ωφελήσει τους πλούσιους, ενώ η οικονομική κρίση ουσιαστικά έπληξε τους πλέον φτωχούς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η προπαρασκευαστική συνάντηση αυτή την εβδομάδα και είδαμε ποια ήταν οι συνέπειε ε, τη ποσοτική χαλάρωση του ΕΚΤ για περίοδο τριών μηνών. Και έγινε μία διαπίστωση ότι έγινε μία μεταφορά μεταξύ γενναιών Οι πιο ηλικιωμένοι γίνονται πιο πλούσιοι και πιο φτωχοί γίνονται οι πιο νέοι και αυξάνονται οι ανισότητες. Είπατε λοιπόν στα εισαγωγικά σας σχόλια ότι η ρευστότητα από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. Δεν το βλέπουμε αυτό όμω στην πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν τεκμήρια, να φτάνουν τα χρήματα αυτά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στεγνώσει με την οικονομική κρίση. Έχω λοιπόν μια πρόταση να σα κάνω, να ακούσω ποια θα ήταν η απάντησή σα σε αυτήν. Την Τετάρτη θα ξεκινήσω μια έκθεση για το πράσινη ποσοτική χαλάρωση, για να χρησιμοποιείται η χαλάρωση με στρατηγικό τρόπο, για να μπορούν να, χρησιμοποιούνται πράσινα ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό θα σήμερα θα, θα, πρέπει να δαπανηθούν καινούργια χρήματα για ανανεώσιμες, ε, για μόνωση, για πράσινους σκοπούς, για να δοθεί μια όθηση με στρατηγικό τρόπο για να υπάρξει αυτή η μετάβαση. Πώς σας φαίνεται λοιπόν η ιδέα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω την απάντηση σε δύο τμήματα. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω μία απόχρωση σε ό,τι αφορά το σχόλιο που, έκατε, που κάνατε για την έλλειψη διοχέτευσης των χρημάτων αυτών στην πραγματική αγορά και για τις ανισότητες που προκαλούνται. βλέπουμε πραγματικά να υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία τυχετεύονται στην αγορά. Με πάσα ειλικρίνεια βλέπουμε ότι τράπεζες και άλλοι επενδυτέ ή ασφαλιστικές πολλούν τα ομόλογα του και βλέπουμε και οι τράπεζες να αυξάνουν τα δανεισμούς και οι ασφαλιστικές και άλλοι μακροπροθεσμοί επενδυτές να κινούνται πιο, προς πιο επικίνδυνες επενδύσεις υπό την έννοια ότι σχετίζονται πιο πολύ στην πραγματική εικόνα με την πραγματική οικονομία και δεν είναι μόνο κρατικά ομόλογα. Αυτό λοιπόν το παρατηρούμε. Επίσης παρατηρούμε μία ε, αναδιάρθρωση των ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι ανακάμπτει η ευρωπαϊκή οικονομία. Με μία ισχύ που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι η ανάκαμψη αυτή είναι μέτρια ακόμα. Είναι πιο ευρία όμως και κινείται και προέρχεται από την κατανάλωση, από τις επενδύσεις όπως είπα και προηγουμένως και προσφάτως δε και από τις εξαγωγές. Η ανάκαμψη λοιπόν αυτή προκαλείται σίγουρα από την νομισματική μας πολιτική, αλλά θα έπρεπε να διευκρινίσω και από άλλους παράγοντες. Από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, για παράδειγμα. Υπάρχει όμως. Δεν είμαι τόσο πεπισμένος, λοιπόν, ότι η νομισματική μας πολιτική δεν ε, επικοινωνεί με την πραγματική οικονομία. Και αυτό για τον εξή λόγο. Σε αντίθεση με το 2012, τώρα το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη στην ζώνη του ευρώ είναι πολύ πιο υγιές και στεναρό, γιατί οι τράπεζες αυτές περάσανε την συνεκτική αξιολόγηση και επίσης περάσανε από το check-up, αν θέλετε, από τον έλεγχο των ισολογισμών τους και πλέον είναι σε πολύ καλύτερη θέση να διαβιβάσουν αυτές τα, αυτά τα κίνητρα στην πραγματική οικονομία. Άρα, τα επιτόκια δανεισμού πέφτουν. Το διαπιστώσαμε αυτό Επίσης, πιο σημαντικό, έχουμε τα αποτελέσματα δύο ερευνών, δύο ε, αξιολογήσεων για τον δανεισμό των τραπεζών η μία, η οποία γίνεται από την Ευρωπαϊκή Διαδική Τράπεζα και ζητά από διάφορες τράπεζες να αξιολογήσουν το επίπεδο πιστώσεων, κατά πόσον δανείζουν πιο πολύ ή πιο λίγο σε σχέση με το παρελθόν και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αλλαγή. Οι απαντήσεις λοιπόν οι οποίες λάβαμε στα πλαίσια της μελέτης είναι ότι έχουν βελτιωθεί τα επίπεδα δανεισμού και δεν δανείζουν τόσο πολλοί τράπεζες πλέον βάσει της αντίληψης του κινδύνου, δηλαδή δεν αρνούνται δάνεια λόγω ρίσκου, αυτός ο παράγοντας έχει εκλείψει και ούτε ο καθεξής σε ό,τι αφορά την πλευρά των τραπεζών. Άλλη μια έρευνα που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Διεκτική Τράπεζα, αν δεν κάνω λάθο, όπου υπάρχει μεγάλη δειγματοληψία πολλών ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερωτούνται κατά πόσον, πώς αξιολογούν την, ε, τις πιστώσεις που λαμβάνουν. Είναι ενθαρρυντικές οι απαντήσεις. Δεν λέω ότι αυτό αποτελεί απόρρια μόνο τη προσωπικής χαλάρωση. Ενδεχομένω, ενδεχομένως να αποτελεί και το αποτέλεσμα των προηγούμενων νομισματικών μέτρων που είχαμε λάβει. Αλλά εν γέννη διαπιστώνουμε Χρειάζομαι πιο πολύ χρόνο, Πρόεδρε. Ναι, Πρόεδρε, αφήστε τον να απαντήσει στην ερώτηση που έκανα, συγκεκριμένη ερώτηση που έκανα. Ναι, ναι χρειάζομαι πιο πολύ χρόνο, Πρόεδρε. Η ΕΚΤ, λοιπόν, δεν μπορεί να αγοράσει άμεσα α, ομόλογα από την Τράπεζα Επενδύσεων. Και γι' αυτό το λόγο απάντησα όπως απάντησα στις τελευταίες δύο Θα υπάρξει ε, χρηματοδότηση, νομισματική χρηματοδότηση μας παρουσιάσετε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα ομόλογα, θα πρέπει να ε, πληρούν τους όρους ε, αξιολόγησης. Και στην περίπτωση αυτή σίγουρα θα μπορέσει να τα αγοράσει τα ομόλογα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η Ευρώπη και το ευρώ, και η Ευρώπη το αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διχοτομημένη κατά κάποιο τρόπο κατάσταση. Φαίνεται παράδοξο μια χώρα όπως ε, η ε, Ελλάδα έχει ας πούμε την, τη, τη στάση πληρωμών πάνω από το κεφάλι της για ένα δις ενώ η τράπεζα της Φραγκφούρτης έχει δυνατότητες μέχρι τρία δις. Επίσης δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει και παρά μόνο για τις ε, τράπεζες. Ε, να υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία που έχουν τεράστιο ε, πλεόνασμα σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη κατάσταση στην, Νότια Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να, ακολουθούμε όλοι ένα, πρότυπο σαν αυτό που δημιούργησε στο Λουξεμβούργο ο πρόεδρος Γιούνκερ ή σαν τα άλλα αλλά τα οποία αποκάλυψε ο Φαλσιάνη ε, και από την άλλη πλευρά ε, να ε, έχουμε την Ευρώπη η οποία με δάκρυα και αίμα προσπαθεί να επιβιώσει το ένα κομμάτι της Ευρώπης ενώ το άλλο είναι πλούσιο και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσείς κύριε Ντράγκη πραγματικά δουλεύετε από ό,τι φαίνεται μονάχα για αυτούς που κρύβονται πίσω από τις οθόνες τους και περιμένουν μία λέξη σας έτσι ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν πουλήσουν ή να αγοράσουν ε, και ε, επομένως ε, να ε, ε, προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν. Δεν είναι δυνατόν ε, να μην λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία αυτά τα οικονομικά τα οποία δείχνουν ακριβώς ότι μονάχα το τροπεζικό σύστημα δίνει χρήματα και δανείζει χρήματα σε αυτούς που είναι ήδη πλούσιοι σε αυτούς ή σε αυτούς που τους ζητάνε να βάλουν ακόμα και το κεφάλι τους που λέει ο λόγος σαν εχέγγυο. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία να είναι η Ευρώπη τη σούπερ έκπτωση να είναι η Ευρώπη Ευρώπη όπου οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Ίσως τώρα είναι η δικιά σας ευκαιρία κύριε Δράγκη έτσι ώστε να καταλάβετε Πώς ζει ο κόσμος. Και εδώ έρχεται η ερώτησή μου. Είναι δυνατόν ε, να μην ε, μπορείτε να καταλάβετε ε, ότι, δεν, ότι πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ θαραλέες. Ο Γιούγκερ με τον Τούσκο και μαζί σας να πάρουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες να δημιουργήσουν ένα ικανοποιητικό φορολογικό καθεστώς. Να, να, να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι στο κέντρο και όχι οι κερδοσκόποι στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας. Ε, ε, κοιτάξτε, ε, στην Ευρώπη, το είπα και στην αρχή, τα πράγματα είναι διχοτομημένα. Αυτά που πρέπει να κάνετε με την Ελλάδα, αυτά που πρέπει ενδεχομένως να κάνετε με το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πρέπει να τα κάνετε τώρα. Ε, now the answer... Η απάντηση είναι, πρώτα απ' όλα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, οι τράπεζες και οι αγορές υπάρχουν και είναι η μόνη διάβλη που έχουμε για την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία. Κάποιες από αυτές τις πολιτικές μπορεί να αυξήσουν την ανισότητα από τη μία πλευρά, αλλά συγχρόνως ας σκεφτούμε ποια είναι η κύρια πηγή της ανισότητας, είναι η ανεργία. Στο βαθμό που αυτές οι πολιτικές βοηθούν και πράγματι βοηθούν να ανακάμψει η απασχόληση, μειώνουν την, την ανισότητα. Είναι καλύτερη μια τέτοια πολιτική λοιπόν η οποία είναι επεκτατική από μια πολιτική η οποία είναι περιοριστική σε αυτή την χρονική στιγμή. Θέλετε να αυξήσουμε τα επιτόκια λοιπόν όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Αυτό ζητάτε. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Από αυτή την άποψη πιστεύουμε και πράγματι βλέπουμε να βελτιώνεται η πραγματική οικονομία. Γι' αυτό ακολουθούμε το δρόμο αυτό γιατί είναι ο καλύτερος δρόμος για να μειώσουμε τις ανισότητες. Για το άλλο ερώτημα, γιατί δεν ερχόμαστε σε συμφωνία με τους άλλους. Συγγνώμη. Υπάρχει έκθεση των τεσσάρων προέδρων. <clears throat> Για πρώτη φορά γίνεται αυτή η προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι απόψεις διαφορετικών θεσμικών οργάνων και επίσης άλλων φορέων. Δηλαδή να έρθουν από κοινού όλες οι απόψεις αυτών που βρίσκονται στο επίκεντρο <clears throat> της αντιμετώπισης της τωρινής κρίσης. Ήταν αρκετά επιτυχής προσπάθειες των τεσσάρων πρόεδρων στο παρελθόν, γιατί τα πορίσματα αυτής της έκθεσης έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οδήγησαν προς την Τραπεζική Ένωση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχετε περιγράψει. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα αυτά. Δεν τα, ανα, δεν τα ανακαλύπτουμε σήμερα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και τουλάχιστον θα έχουμε προσπαθήσει, έστω και αν δεν έχουμε επιτύχει ε, μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπερνάν Μωρό. Κύριε Πρόεδρο, καλημέρα σας. Για το θέμα της Ελλάδος. Η Τρόικα εξακολουθεί να έχει ένα ψυχότραμα με την ελληνική κυβέρνηση για να ασκήσει την πίεση στην κυβέρνηση Τσίπρας και να πιέσει την ελληνική κοινωνία σε μια αυστηρή λιτότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή το σύστημα Target 2 του ευρωσυστήματος εξασφαλίζει ότι επαναπληρώνεται το ελληνικό δάνειο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί λοιπόν να μην συνεχίσετε τη χρηματοδότησή σας με την έκτακτη χρηματοδοτική αρρωγή ρευστότητος προς την Ελλάδα. Και επίσης για το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Εμείς υποστηρίζουμε το να υπάρχει παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά με την, υπο, με την ε, προϋπόθεση ότι αυτό οδηγεί σε αποπληρωμή των χρέων. Ενώ εδώ δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε να χρηματοδοτούνται μονάχα οι ιδιωτικέ τράπεζες και οι αγορές κεφαλαίων, αλλά δεν χρηματοδοτείται η παραγωγική οικονομία και δεν γίνεται τίποτα για την ε, απασχόληση. Πάρα πολλοί έχουν εποφεληθεί από αυτές τις ενέργειες με, την, ε, με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Εσείς λοιπόν, σε τεχνικό επίπεδο, θα ήσασταν έτοιμος να προχωρήσετε σε μία τροποποίηση του άρθρου 123 ώστε να μπορείτε να χρηματοδοτείτε κατευθείαν το ε, κρατικό χρέος για να υπάρξει σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ. Και τέλος, δεοντολογία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να επανέλθω στην δήλωση του κ. Μπενουά Κέρε που κατά τη δική μου άποψη είναι μια σοβαρή υπόθεση. Απαντώντας σε ορισμένου επενδυτές, ο κύριος Κερέ είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τις αγορές αξιογράφων μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι μειώθηκαν αμέσως τα ε, επιτόκια και αυξήθηκε η αγορά των μετοχών και μειώθηκε η ισοτιμία του ευρώ. Αυτοί λοιπόν που είχαν πρώτη την πληροφορία αυτή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να αξιολογήσουν μια προνομιακή πληροφόρηση. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο το οποίο πρέπει να οδηγήσει σε ανάληψη δράση από την Κεντρική Τράπεζα. Θα γίνει μια πειθαρχική ή μια δικαστική έρευνα εναντίον του κύριου Κέρα για να διευκρινιστεί αυτή η κατάσταση. Θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα σφάλμα, για ε, μια άδικη πράξη του ε, κυρίου Κέρα που αξίζει κυρώσει για αυτό το λόγο. Να είμαι σύντομο απαντώντας στο ερώτημα αυτό και θα είμαι κάπω πιο μακροσκελής στο δεύτερο ερώτημα για το πρώτο ερώτημα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικέ απόψει σε σχέση με τι συνθήκε, αλλά δεν είναι δικό μα εγχείρημα να αλλάξουμε την συνθήκη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει από τι κυβερνήσει. Είναι κάτι το οποίο εναπόκειται σε εκλεγμένου νομοθέτε. Δεν είναι το έργο θεσμικών οργάνων. Για το δεύτερο ερώτημα. Για να αντιμετωπίσω πολύ προσεκτικά αυτό το υποτιθέμενο σκάνδαλο που αναφέρατε για τον κύριο Κιωρέ. Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα και καταρχήν για να διαλύσω όλες τις παρεξηγήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε. Ο κύριος Κερέ είπε ότι, παραθέτω, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εποχιακές στάσεις στην αγορά με μια ιδιαίτερη περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι τα μέσα Αυγούστου που έχει χαμηλότερη ρευστότητα στην αγορά. Το ευρωσύστημα λαμβάνει αυτό υπόψη στην εφαρμογή του προγράμματός του για τη διευρυμένη αγορά αξιογράφων με το να εμπροστοφορτήσει τις αγορές του τον Ιούνιο για τα αξιόγραφα. Επί τη βάση των στοιχείων που καλύπτουν το πρώτο τμήμα του Μαΐου, όπως έχουν αναφερθεί στις εβδομαδιαίες ανακοινώσεις της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ιστοσελίδα της και που δημοσιεύτηκαν στις 11 ε, και 18 Μαΐου 2015, δηλαδή πριν από την ομιλία του κυρίου Κέρε στο Λονδίνο, η αγορά της εμπροστοφόρτησης των αγορών είχε αναφερθεί ήδη με ένα τρόπο πάρα πολύ σαφή σε αυτές τις ανακοινώσεις. Και αυτό δεν οδήγησε σε καμία επιτάχυνση αγορών στο δεύτερο τμήμα του Μαΐου έναντι των προηγουμένων αγορών. Επομένως, μια μετριοπαθής μπροστοφόρτιση, δηλαδή μια μικρή τροποποίηση των αγορών για να μην υπάρξουν εντάσεις στην αγορά τον Αύγουστο, Φυσικά αυτό δεν αποτελεί καμία αλλαγή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επομένως δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως μια ανακοίνωση αλλαγής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Περαιτέρω, όπως είπα και στην επιστολή στην κυρία O'Reilly, την ε, διαμεσολαβήτρια, η ομιλία αυτή επρόκειτο να δημοσιευτεί το βράδυ της ομιλίας στην ιστοσελίδα μας, αλλά δημοσιεύτηκε μόνο το επόμενο πρωί λόγω ενός σφάλματος, μιας εσωτερικής αποτυχίας επικοινωνίας κατά την διάρκεια της ε, δημοσίευσης, γιατί η ομιλία έγινε εκτός του ωραρίου εργασίας. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αναθεωρήσει τις διαδικασίες της ώστε να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο σφάλμα. Θα υπάρχουν περαιτέρω έλεγχοι εσωτερικά και διασταυρούμενοι έλεγχοι για να εξασφαλίσετε ότι γίνεται η έγκαιρη δημοσίευση αυτών των δηλώσεων σε όλες τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σταντελάνε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας ε, εξηγείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας για διάφορα ε, σημεία κλειδιά και θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα του πληθωρισμού και αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά τις ε, προσδοκίες αύξησης μετριοπαθού αύξηση, κοιτώντα και τα γερμανικά ομόλογα και τι εξελίξει του, η μείωση τη αξία του τελευταία. Είπατε ότι υπάρχει μεγάλη αστάθεια και διακύμανση για να το εξηγήσετε αυτό όλοι, όμω γνωρίζουμε ότι ενδεχομένω να αποτελεί αυτό ένδειξη ε, προσδοκία μεγαλύτερου πληθωρισμού των αγορών στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν και αυτό ο παράγοντα πέρα από την διακύμανση. Και περνάω λοιπόν έτσι στην ποσοτική χαλάρωση και στο ερώτημά μα. Είπατε με σαφήνεια ότι σκοπεύετε να συνεχίσετε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Τι θα γίνει με τις προσδοκίες της αγοράς αν επαληθευτούν, αν υπάρχει πιο γρήγορη αύξηση του πληθωρισμού. Θα συνεχίσετε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 ακόμα και ένα πληθωρισμός φτάσει στο 2% και σε ποιο σημείο προβλέπετε να σταματήσετε ο πληθωρισμός, μιας και αποτελεί το βασικό σας στόχο, αποτελεί το μοναδικό λόγο, την μοναδική αιτία για την ποσοτική χαλάρωση, την επίτευξη του 2%. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι ή ίσως άλλες ε, παράπλευρες ε, συνέπειες ε, από την ποσοτική χαλάρωση που ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ επωφελείς και ενδεχομένως να δικαιολογήσουν τη συνέχιση του προγράμματος, ακόμα και αν δεν χρειάζεται για τον πληθωρισμό καθεαυτό. Σας ευχαριστώ. Μπορεί κανείς να φανταστεί διαφόρους λόγους για τους οποίους ε, έγινε αυτή η αύξηση στις, ε, στα κρατικά ομόλογα. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι η προσδοκία αύξησης πληθωρισμού. Ένας από τους πολλούς λόγους που έχουμε ακούσει τελευταία. Αν αυτό ίσχυε ωστόσο, θα σήμαινε ασφαλώς αυτό ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι πολύ επιτυχής και οι αγορές προβλέπουν ακριβώς ότι θα πετύχουμε το στόχο αυτό. Επίσης, αν το πρόγραμμα που υποτίθεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι το 2016 θεωρηθεί υπερβολικό από τις αγορές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προβλέπουν μεγαλύτερη επιτυχία από ότι εμείς οι ίδιοι σε ό,τι αφορά την ποσοτική χαλάρωση. Όπως και να έχει, στην παρούσα φάση πιστεύουμε ότι το, η επίτευξη του στόχου μας το 2016 και το 2017 με το 1,8% να εξαρτάται απόλυτα από την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, όπως έχει σχεδιαστεί. Με άλλα λόγια, προβλέπουμε αυτό το υψηλότερο πληθωρισμό για τα επόμενα δύο χρόνια, μόνο και μόνο επειδή βασιζόμαστε στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Ρωτήσατε κατά πόσο το κάνουμε αυτό για το μοναδικό σκοπό της σταθερότητας των τιμών. Ναι, μας περιορίζει η εντολή μας. Η εντολή μας μιλάει μόνο για σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, και αυτό νομίζω καταδεικνύει ότι είναι πολύ πιο ευρύ στόχος αυτή η σταθεροποίηση και η σταθερότητα των τιμών. Προσπαθώντα να πετύχουμε λοιπόν τη σταθερότητα των τιμών, γνωρίζουμε ότι υπάρχει η κοινή νομισματική πολιτική μας που επηρεάζει με θετικό τρόπο την ανεργία βοηθά να μειωθεί το χάσμα και υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη. Άρα υπό την έννοια αυτή η επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών συνοδεύεται με στόχους που σχετίζονται πιο άμεσα με την πραγματική πλευρά της οικονομίας. Σας ευχαριστούμε. Ο κ. Φον Φάιτσέκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Δράγκη, πάντα τιμή και χαρά να σα ακούμε. Παρά το γεγονό ότι δεν επεκτάθηκατε για το μέλλον ε, τη Ευρωζώνη, Μία ερώτηση για την Ελλάδα, φοβάμαι, και για την οργάνωσή σας ε, ως μία οργάνωση που βασίζεται σε κανόνες. Αν η Ελλάδα σταματήσει να εξυπηρετεί τους ε, διεθνείς πιστωτές τους, θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα συμβαίνει με το πρόγραμμα αρρωγή ρευστότητα για τι ελληνικέ τράπεζε. Και συγκεκριμένα, ποια θα είναι η νομική βάση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τερματίσει την έκτακτη ε, αρρωγή ρευστότητα δεδομένου του γεγονότο αυτού. Επειδή οι ελληνικέ τράπεζε έχουν μεγάλη έκθεση σε ε, ομόλογα σύντομη ε, και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι θα έπρεπε να γίνει για, το, για να αυξηθεί το κούρεμα του εθνικού χρέους της Ελλάδας και πώς μπορεί να υπάρξει η διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμης ή μακρυπρόθεσμης οριμότητας. Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για την ε, προοπτική δανεισμού της Ελλάδας ο μηχανισμό σταθερότητα. Thank you. Ε, Let Σας ευχαριστώ. Να σας απαντήσω γενικά. Δεν θέλω να αποδηθώ σε εικασίες. Σε περίπτωση από, την, ε, από τα λόγια των Ελλήνων ηγετών ξέρουμε ότι οι πληρωμές αυτές θα πληρωθούν εγκαίρως και 100%. Ε, Άρα δεν έχει νόημα να εικάσω το τι θα κάναμε σε περίπτωση που θα υπήρχε στάση πληρωμών στην παρούσα φάση. το δεύτερο σημείο που θίξατε για τον ε, έκπληκτη αρρωγή ρευστότητα και πώς ε, λειτουργεί η διαδικασία λήψης ε, αποφάσεων. Πρόκειται για μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας. Δεν είναι απόφαση του, του, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας. Γίνεται το αίτημα έγκρισης αύξησης του ELA Προ τι ελληνικέ τράπεζε στην προκειμένη περίπτωση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μόνο να απορρίψει το έτοιμο αυτό με πλειοψηφία δύο τρίτων. Και αυτό γιατί όταν σχεδιάστηκε η εκδιαρρογή ρευστότητα στι αρχέ τη Οικονομικής Ένωση, υπήρχε η αντίληψη ότι θα έπρεπε κανεί να διατηρήσει κάποιες από τις ε, αρμοδιότητες των εθνικών κρατικών τραπεζών. Δεν υπήρχε ιδέα του επόπτη τότε. Άρα, η ιδέα ότι θα υπήρχαν αφαιρέγγιες τράπεζες σε μια χώρα και ότι αυτές οι τράπεζες θα έπρεπε να επηρεάζονται πιο πολύ από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, ήταν αυτή που επικρατούσε τόσο. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίοδο οφείλονται αυτά που ισχύουν. Είναι σημαντικό όμως να θυμόμαστε ότι δεν πρόκειται για απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ειδικής πλειοψηφία για να υπάρχει απόρριψη της πρότασης του ELA. Το θέμα για την Ελλάδα και τον δανεισμό από το Μηχανισμό Σταθερότητας προκειμένου να αγοραστούν αυτά τα ομόλογα από το Μηχανισμό Σταθερότητας είναι κάτι το οποίο συζητάτε. Δεν είμαι βέβαιος και εδώ θα πρέπει να επιτύξω ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είμαι βέβαιος ότι η παρούσα συνθήκη του μηχανισμού σταθερότητας επιτρέπει αυτή την δυνατότητα. Αλλά εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτά που σας λέω. Του τουλεχθέντος δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να επιληθεί πρόγραμμα για την αγορά αξιογράφων ε, στην αγορά. Υπάρχουν άλλοι οδοί. Είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση να εστιαστούμε στις βασικές απαιτήσεις για την επίτευξη συμφωνίας και όχι τόσο στις ε, τεχνικές λεπτομέρειες της χρηματοοικονομικής φύσεως που θα μεταφράσουν αυτή τη συμφωνία. Και ουσιαστικά έχουμε δύο κατηγορίες στόχους. Να περάσουμε σε μια συμφωνία, να φτάσουμε σε μια συμφωνία για τα μέτρα πολιτικής τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στην Ελλάδα και προκειμένου αυτή η συμφωνία να αποτελέσει βάση της απόφασης των μελών του Eurogroup. Αν τα μέλη του Eurogroup αποφασίσουν θετικά βάσει της συμφωνίας αυτής σε επίπεδο τεχνικών, τότε οι διατάξεις για τις επόμενες 12 μήνες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και οι εκταμιεύσεις και ε, ένα μεγάλο τμήμα των εκταμιεύσεων αυτών θα είναι χρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 16 δις από τα 21, αν δεν κάνω λάθος αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δηλώνει ότι μπορεί να απελευθερώσει τα χρήματα αυτά μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς εγγυήσει για τη χρηματοδότηση του επόμενου προγράμματος. Και αυτό επειδή πιστεύουν και νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι θεσμοί για την αξιολόγηση αυτή ότι χρειάζεται και περαιτέρω χρηματοδότηση. Και αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη κατηγορία όρων. Τα κρατημέλη θα πρέπει να επιλύσουν το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση προκειμένου το Διεθνές Δημοκρατικό Ταμείο να μπορέσει να δώσει σήμερα. Τι δώσει. Δεν είναι απλό, δεν είναι απλό, το φαντάζεστε, αλλά είναι απαραίτητο. Αυτές λοιπόν οι δύο κατηγορίες ε, όρων θα πρέπει να συντρέχουν. Thank Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Είναι, λοιπόν, και ευθύνη των κρατών μελών και της ελληνικής πλευράς. Ο Μάρκος Φέρμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Δύο σύντομα ερωτήματα έχω να σας θέσω. Πρώτα, σε σχέση με την ποσοτική χαλάρωση. Είπατε προηγουμένως σε μια ομιλία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι αυτή η πολιτική μπορεί να λειτουργήσει μονάχα σε συνδυασμό με πολιτικά μέτρα τα οποία πρέπει να, είναι, να συνάδουν ώστε να λειτουργήσει, να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα και να δημιουργηθούν και οι απαραίτητες δομές. Και ότι δεν υπάρχει πάντα αυτό το μείγμα προϋποθέσεων σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν εφαρμόσει αυτό το σύστημα της πολιτικής χαλάρωσης. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η δράση, πώς θα μπορέσετε να επιτύχετε αυτό που θέλετε και μήπως θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, να μειώσετε την πίεση για μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Και το δεύτερο θέμα, για την ε, υποστήριξη με την το έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ελληνικής τράπεζας. Η πρόεδρος του μηχανισμού επίλυσης τραπεζών είπε ότι αυτό οδηγεί σε μια υφέρπουσα διαδικασία ε, αφαιρεγγιότητος των τραπεζών. Πώς εσείς ε, κρίνετε αυτή την άποψη της κυρίας Κιόνικ που είναι η επικεφαλής του μηχανισμού επίλυσης τραπεζών. Well, uh, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σχολιάσω τα ε, δηλαθέντα από την κυρία Κένιγκ. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω τι μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική και τι δεν μπορεί να κάνει. Η νομισματική πολιτική μπορεί να βοηθήσει ε, στην κυκλική ανάκαμψη, δηλαδή μία ανάκαμψη για τα επόμενα δύο χρόνια, μία ανάκαμψη, όπου ας πούμε τα κυκλικά συστατικά της ανεργίας ας πούμε θα αντιμετωπιστούν και ενδεχομένως ευελπιστούμε ότι θα εξαφανιστούν. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν δεν είναι δυνατόν παρά μόνο μέσα από κάποιες ε, έμεσες ας πούμε πράξεις δεν μπορεί να οδηγήσει ε, σε διαρθρωτική ανάκαμψη. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα ολοκληρωθεί η κυκλική επίπτωση της νομιωτικής πολιτικής ε, και αν τότε δεν έχει υπάρξει θετική ε, ανάκαμψη ας πούμε στην διαρθρωτική ε, φάση τότε θα χρειαστεί μια φάση σταθερότητας τιμών ή τα, τα προβλήματα, θα πρέπει να καλυφθούν τα επιπλέον προβλήματα σταθερότητας τιμών τα οποία δεν θα έχουν επιτευχθεί μέχρι τότε και αυτά μπορούν να καλυφθούν μονάχα από τη λεγόμενη δημοτική πολιτική και όχι από την νομισματική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν συχνά επαναλαμβάνω ότι εάν θέλουμε η νομισματική πολιτική να οδηγήσει σε πλήρη ανάκαμψη θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από φιλόδοξο ε, διαρθρωτικό πρόγραμμα να μην λησμονούμε όταν βλέπουμε ας πούμε τα ποσοστά της ανεργίας έχει ξεπεράσει τώρα το ποσοστό αυτό το 11% σε μέσο όρο στην Ευρωζώνη ε, αλλά αυτό κρύβει τις ε, τεράστιες διαφορές ε, των εθνικών στοιχείων που αφορούν τα ποσοστά ανεργίας αλλά εάν δούμε τα χρόνια πριν από την κρίση ας πούμε το 2007 νομίζετε ότι πραγματικά τα ποσοστά ήταν πολύ χαμηλότερα. Όχι, ήταν περίπου 9% ο μέσος όρος. 9% και μάλιστα το ποσοστό αυτό διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, εντάξει ναι, περίπου 9% για πολλά χρόνια, όταν οι κυκλικές πολιτικές άλλαζαν, δεν ήταν ίδιες. Ας πούμε, για πολλές ε, χώρες Δέκα χρόνια πριν από την κρίση ε, ήταν χώρες ε, όπου αυξήθηκαν ε, οι κρατικές δαπάνες ακολουθούμενες και από σημαντικέ αυξήσεις των φορολογικών εσόδων με ταυτόχρονες πολλές περικοπές των δαπανών. Ωστόσο, και πέρα από αυτές τις ε, ε, μεγάλες ε, περικοπές των κρατικών ταπανών δεν είδαμε τρομερή αύξηση της ανεργίας παντού. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση της ελεύθερης αγοράς και αυτό μπορεί να ισχύει και ίσως και περισσότερο μάλιστα στην αγορά των προϊόντων, αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση, σε, συγγνώμη, στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτού του είδους τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν από, στρατι... Ε, από διαρθρωτικές ε, πολιτικές και όχι από νομισματικές ε, πολιτικές μάλιστα. Σε περίπτωση που κινηθούμε προς την ανάκαμψη της αγοράς υπηρεσιών, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις εγγενείς ανισορροπίες της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Κύριος Φερνάντης Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δράγκη για την απάντηση, την έγγραφη απάντηση που έδωσε στο ερώτημα που είχα διατυπώσει εγώ προς αυτό στην Επιτροπή μας και σήμερα θα ήθελα να κάνω το σχόλιο το εξή ότι βάσει των πληροφοριών που ε, έχει δοθεί στο Κοινοβούλιο μας, πέντε από τα κράτη-μέλη που ακόμα δεν είναι, δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης θα μπορούσαν να τηρήσουν τις προϋποθέσεις για να μπουν στον μηχανισμό ισοτιμιών 2 και να προχωρήσουν προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Βουλγαρία, Ρουμανία, Σουηδία, Πολωνία. Είναι έτοιμες αυτές οι πέντε χώρες λοιπόν. Μπορούν λοιπόν να μπουν στην Ευρωπαϊκή ε, οικονομική και Νομισματική Ζώνη εάν κάνουν την απαραίτητη πολιτική απόφαση. Το άρθρο 119 της Συνδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εργαστούν για να τηρήσουν τους κανόνες σύγκλησης και εν καιρό να ζητήσουν την ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ. Τους τελευταίους μήνες συζητάμε πολύ για το πώς θα βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Εσείς μιλήσατε για την έκθεση των πέντε προέδρων που περιμένουμε τη δημοσίευσή της και τονίσατε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα κβαντικό άλμα, ένα ποιοτικό άλμα στην αρχιτεκτονική διακυβέρνησή της. Θα ήθελα όμως να ακούσω μεγαλύτερη επιμονή από τη δική σας πλευρά, ώστε οι χώρε αυτές που έχουν την νομική υποχρέωση να μπουν στη ζώνη του ευρώ, εκτός από τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και τηρούν τα κριτήρια, να κάνουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να μπουν στην ε, ζώνη του ευρώ για να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στην Τραπεζική Ένωση, στην Κεφαλαιακή Ένωση και φυσικά και στη μεγαλύτερη δημοκρατική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να αφορά, πρέπει να διέπει όλες τις χώρες που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ και όχι μερικές μόνο από αυτέ. Ευχαριστώ, λέω κύριο κύριος αν γυρίσουμε τρία ή τέσσερα χρόνια πίσω στο χρόνο, είδαμε ότι κάποιες χώρες μπήκανε στη ζώνη του ευρώ και άλλες χώρες που ήταν εξίσου αποφασισμένες και έλεγαν ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο ευρώ. Παρά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές που αναφέρατε είναι μέσα στα οικονομικά κριτήρια σύγκλησης για τη ζώνη του ευρώ, η πολιτική τους θέληση δεν υπάρχει ή δεν έχει οριμάσει αρκετά για να φτάσει στο στάδιο που θα θέλανε να μπουν πράγματι στη ζώνη του ευρώ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούμε. Είναι μια πολιτική θέληση που πρέπει να την αποδεχτούμε. Αρχικά θεωρήσαμε ότι όσο ευρύτερη είναι η νομισματική ένωση τόσο καλύτερα. Αυτή ήταν η φιλοδοξία μας. Σήμερα όμως αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του να δαπανούμε την προσπάθειά μας προς την κατεύθυνση της διεύνησης της Ένωσης, της Νομισματικής Ένωσης ή του να, χρησιμοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να την ενισχύσουμε, να έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση στον δημοσιονομικό τομέα και στον πολιτικό τομέα, εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παύλος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. στο θέμα της Ελλάδος. Ο κύριος Βαρουφάκης τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, του ελληνικού χρέους. Ποια είναι η απόψή σα για την αναδιάρθρωση του χρέους. Είναι μια προτεραιότητα ή όχι. Λαμβάνοντας υπόψη του ότι το επίπεδο των ε, τόκων που πληρώνει η Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από αυτό που πληρώνουν άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Και αντίθετα, κατά την άποψή σα, μήπω θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα η ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτέ θα πρέπει να οδηγήσουν στι μεταρρυθμίσεις, ακόμα και αν βραχεί πρόθεσμα έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Μήπω θα ήταν λοιπόν πιο πρόσφορο για την ελληνική κυβέρνηση, αντί να έχει αυτή η μονομανία με την αναδιάρθρωση του χρέους της, να προσπαθήσει να βρει μια λύση για τον αντικό αντάκτυπο, αντίκτυπο που θα έχουν οι βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις με στόχο να επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και επίσης απαντώντας στην κυρία Φερέιρα, είπατε ότι στην περίπτωση ενός γεγονότος το οποίο κανείς δεν θα ήθελε αλλά θα μπορούσε να προκύψει με απρόβλεπτο τρόπο, θα πρέπει να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα για να έχουμε μια πιο ισχυρή οικονομική και νομισματική ένωση και μια πολιτική ένωση. Είναι γεγονό ότι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά συγχρόνω εσείς, όπως κάνατε και το 2012, μπορείτε να δώσετε περισσότερο χρόνο ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Στην υποθετική περίπτωση, μακάρι να μην γίνει ποτέ, κάποιο τέτοιο απρόβλεπτο γεγονός. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δώσει περισσότερο χρόνο στα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το απαραίτητο ποιοτικό άλμα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Δράγκη. Να σας πω. Δεν θέλω να πάρω θέση ε, σχετικά με το εάν χρειάζεται το ένα ή το άλλο πράγμα, γιατί δεν ε, αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Ε, ε όσον αφορά το δάνειο EFSF, έχει 0,5% ε, ε, ε, της επιτόκιο. Η δε μέση ορίμανση είναι 30 χρόνια και επομένως καταλαβαίνετε ότι για τα επόμενα 4 χρόνια για την Ελλάδα προκύπτουν υποχρεώσεις περίπου στο μισό από τι άλλες χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται ε, κάπου στη μέση ας πούμε και επομένως ε, τώρα ε, που θα πρέπει να δοθεί η εστίαση αυτό θα πρέπει να το αποφασίσετε εσείς, σίγουρα όχι εγώ. Τώρα η ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Έχω πει επανειλημμένα και θα επαναλάβω ότι θα πρέπει και είναι δυνατόν να υπάρξει μια συμφωνία, μια ισχυρή συμφωνία όπου η ανάπτυξη ε, θα έρχεται παράλληλα με την κοινωνική δικαιοσύνη και με την φορολογική ε, και χρηματοπιστωτική σταθερότητα η βιωσιμότητα, η φορολογική, η δημοσιονομική, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες. Ε, δίνει ε, την υπόσχεση κατά κάποιο τρόπο και θα είμαι εδώ πάρα πολύ γενικός γιατί δεν θέλω να μπω σε εξειδικευμένα στοιχεία του προγράμματος. Δίνει την δυνατότητα εξασφάλισης ενός σταθερού εισοδήματος ας πούμε για τα επόμενα 100 χρόνια. Βεβαίως ενδεχομένως δεν έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο ε, στις ε, τωρινές απαιτήσει. Ε, εάν λοιπόν ο κόσμος δεν καταλάβει, δεν πιστεί ότι μπορεί να ένα μέτρο που προτείνεται ή μια συμφωνία που προτείνεται να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, τότε δεν θα την αποδεχτούν γιατί ε, στην προκείμενη περίπτωση δεν έχουμε τέτοιου είδους λοιπόν ε, δέσμευση για τους ε, κανόνες ή μάλλον είχαμε συχνή αλλαγή των προτινόμενων κανόνων. Αυτό λοιπόν προκάλεσε αστάθεια και πίεση στην ζήτηση. Δεν θέλω να πω πιο συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πάντως σίγουρα ε, θα πρέπει να έχει κανείς και τους τρεις παράγοντες που ανέφερα προηγουμένως έτσι ώστε να επιτευχθεί η νομισματική ε, και η οικονομική σταθερότητα. Το δεύτερο όσον αφορά ε, το κατά πόσο μπορεί να δοθεί περισσότερος χρόνος για αυτό το ποσοτικό άλμα ή εν πάση περιπτώσει ε, για να ε, αλλάξει η διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς ξεχωριστά από μια συνολικότερη νομισματική πολιτική. Το έλεγα και προηγουμένως, η νομισματική πολιτική βοηθάει την κυκλική ανάκαμψη, βοηθάει να ξεπεράσει κανείς κάποια προβλήματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδώσει να, να, να ολοκληρωθεί στο τέλος ε, ε, με μια διαφορετική ε, σημαντική τροποποίηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σανφρεσάντ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η προσωπική χαλάρωση σίγουρα φαίνεται ότι βοηθάει την ανάκαμψη στην ζώνη του ευρώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συχνέ προειδοποιήσει ότι μπορεί να είναι ευαίσθητη και ευάλωτη αυτή η ανάκαμψη και ότι δεν δημιουργεί τόσο θέσεις εργασίας όσο θα χρειαζόταν. Η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα είναι ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ευρωζώνη θα πρέπει να κάνει πιο πολλέ δραστηριότητε αλλαγέ. Αυτό το λέμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά με τη στρατηγική και με τις, τα αποτελέσματα τη παραγωγικότητα δεν είναι επαρκή. Και αυτό έχει μειώσει την ζήτηση στην Ευρωζώνη και έχει καταστήσει πιο δύσκολη τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Μήπω με την τρέχουσα πολιτική ε, οδηγούμαστε σε ένα ε, σταθερό επίπεδο, αλλά όχι στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις αποκλήσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρωζώνης. Δεν σύμφωνείτε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής πριν ε, δοκιμάσουμε οποιοδήποτε τέτοιο κβαντικά άλματα είναι να γίνουν μέτρα για να περιοριστεί και να ανατραπεί ε, αυτές οι αποκλήσεις, οι περιφερειακές αποκλήσεις και να μην αυξηθούν τα χάσματα σε ό,τι αφορά και την ε, σταθερότητα που θέλουμε η απάντηση. Συμφωνώ, συμφωνώ και επαυξάνω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η νομισματική πολιτική μπορεί να βοηθήσει για την κυκλική ανάκαμψη θα βοηθούσε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Όχι. Αυτό θα πρέπει να προκύψει από άλλους παραγοντές, από την εκπαίδευση, τις ικανότητες, τη ανταγωνιστικότητα στην ε, αγορά υπηρεσιών και προϊόντων. Με κρίσιο κατάλογος των ε, παραγόντων που δεν είναι ίδιοι άλλωστε και αναχώρα. Ποικίλουν. Αλλά είναι αυτός καλός λόγος για να αλλάξουμε την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Όχι. Όχι. Γιατί αυτή η πορεία νομισματικής πολιτικής θα μας οδηγήσει στη σταθερότητα των τιμών και όπως ορίσετε, όπως εξήγησα προηγουμένως. Δεν είναι λοιπόν επαρκής αυτός ο λόγος να αλλάξουμε την νομισματική πολιτική. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η νομισματική πολιτική θα αποδώσει 100% τα όσα προσδοκούμε. Όχι μόνο σταθερότητα τιμών, αλλά και χαμηλότερο σταθερά, χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας. Όχι, όχι, όχι, χρειάζονται πολλά ακόμα. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα για να υπάρξει αυτό το άλμα, το κβαντικό άλμα, αυτό το ποσοτικό άλμα ή να επενδύσουμε επειδή δεν έχουμε πετύχει ακόμα βελτίωση στην παραγωγικότητα και στην οικονομική δομή. Έχω την αίσθηση ότι αυτά δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Θα πρέπει να κινηθούμε προς μεγαλύτερη σύγκληση και εκ παραλλήλου θα πρέπει να αναρωτιόμαστε κατά πόσον η, οικονομική, η νομισματική ένωση έχει σχεδιαστεί με στεναρή τρόπο ή όπως σας είπα προηγουμένω κατά πόσον είναι ακόμα ευάλωτη και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες. Είναι σαφές ότι αυτά τα δύο θα πρέπει να κινηθούν παράλληλα. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση και να σχεδιάσουμε μια διαφορετική οικονομική ένωση με χώρες που είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλίνουσες. Εκ παραλλήλου δε, οι χώρες που συγκλίνουν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αδυναμίες ε, της Ένωσης με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Thank you. The last... Ευχαριστώ. Τελευταίος ο ομιλητής είναι ο εισηγητής ε, για το ΕΦΣΙ, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να λάβω το λόγο ενώψη, ενώπιον του Πρόεδρου Ντράγκη. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με την ικανότητα με την οποία κατάφερε να βοηθήσει τον φορέα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να έχει την ακτινοβολία αυτή που έχει σήμερα. Δύο ερωτήματα. Είναι κάποια κράτη-μέλη που έχουν φτάσει σε ένα ιστορικό χαμηλό σε ό,τι αφορά τα, τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. Η χώρα μου έφτασε, η Πορτογαλία έφτασε και σε αρνητικά επιτόκια. Ποιο ήταν ο ρόλος του προγράμματος αγοράς αξιογράφων τη Κεντρική Τράπεζα σε αυτή την εξέλιξη και επίση ποιο ήταν και ο ρόλο, των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει από κάθε κράτος μέλος, ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η επιτεύξη αυτών των χαμηλών επιτοκίων. Δεν έχουμε μιλήσει αρκετά για τις μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που είναι απαραίτητες. Θα ήθελα όμως να θέσω αυτά τα δύο ερωτήματα. Θεωρείτε ότι θα ήταν θετικό ή εφικτό ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο στο ορατό μέλλον, μέλλον ή επίσης αν θα θεωρούσατε σε μεσοπρόθεσμο ή σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να υπάρχει ένας προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ. Νομίζω ότι, ότι το τωρινό επίπεδο επιτοκίων για τα κρατικά ομόλογα στην πλειοψηφία των χωρών της ε, ζώνης του ευρώ, ακόμα και στις χώρες οι οποίες θεωρούνται ότι ήταν χώρες που υπόκειται σε πίεση, είναι κοινό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναλυθεί από τις χώρες αυτές και την επιτυχία των προγραμμάτων που έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις τους και επίσης της παρουσίας τριών παραγόντων των τωρινών συνθήκων της αγοράς, και της ποσοτικής χαλάρωσης. Γενικότερα της ε, νομισματικής πολιτικής που ακολουθείται από εμά. <clears throat> Βέβαια το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο είναι λένε Τα επίπεδα επιτοκίων που έχουμε δει πρόσφατα, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, έχουν αλλάξει βέβαια όπως είδατε. Υπήρξε ανάκαμψη των επιτοκίων με κάποια διακύμανση, αλλά αυτό είναι και κομμάτι της εξήγησης. Αν θέσουμε όμως τον εαυτό μας το ερώτημα, τι είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει σε μόνιμα χαμηλότερο κόστος του χρέους. Η απάντηση είναι λιγότερο η νομισματική πολιτική ή η ποσοτική χαλάρωση. Κάποτε θα τερματιστεί η ποσοτική χαλάρωση. Και τότε για να επιτύχουμε μικρότερο κόστος του χρέους θα πρέπει να στραφούμε στην ικανότητα που θα έχουν μέχρι τότε δημιουργήσει οι χώρες αυτές για να έχουν οικονομική ανάπτυξη, για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Και όπου αυτό είναι απαραίτητο για να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Κάτι ακόμα που πρέπει να σας υπενθυμίσω και δεν πρέπει να το λησμονήσουμε. Η δημοσιονομική παγίωση ένας από τους λόγους για την τωρινή μας ανάκαμψη είναι ότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίσαν οι χώρες μας τα τελευταία χρόνια. Έχουν ξεπεραστεί αυτές οι πιέσεις γιατί υπήρξε μεγάλη πρόοδος για την παγιοποίηση, για την εδραίωση σε την εξυγίανση σε δημοσιονομικό επίπεδο. Μέσω πρόθεσμα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την δημοσιονομική υγεία στην ε, ζώνη του ευρώ, ώστε να μην υπάρχουν πιέσεις προς τα άνω για τα επιτόκια που να προέρχονται από την αντίληψη ότι ορισμένες δημοσιονομικές καταστάσεις δεν είναι βιώσιμε. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή της κρίσης αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα, ότι για πολλά κράτη-μέλη η δημοσιονομική τους στάση θεωρήθηκε από την αγορά ότι δεν ήταν βιώσιμε. δεν ήταν το σύνολο του προβλήματος, αλλά ήταν ένας μεγάλος, ένα μεγάλο τμήμα του προβλήματος. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν και μεσοπρόθεσμα θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ώστε όταν η νομισματική πολιτική έχει εξαντλήσει σε κυκλικό επίπεδο τις επιπτώσεις της, οι οικονομίες σε δημοσιονομικό και διαρθωτικό επίπεδο θα έχουν εξασφαλίσει την ανθεκτικότητά τους και θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν παραγωγικότητα, ανάπτυξη και χαμηλά επιτόκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Άλλη μόνο αυθόρμητη παρέμβαση. Ο κύριο Δράκη δυστυχώ έχει μια άλλη πολύ σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Όλε Λούντβιξον ο πρώτος και ο μόνος που θα δώσω το λόγο. Ε, ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάτε συχνά σε διάφορε περιστάσεις για τις εθνικές μεταρρυθμίσει τις οποίες θεωρούμε ε, χρήσιμες και απαραίτητες προσθήκες της ε, νομισματικής πολιτικής, αλλά παράλληλα μιλάτε για την εξίσωση, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ένα σημαντικό παράγοντα στο θέμα αυτό, στη διάσταση αυτή. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν για την ισότητα αυτή θα πρέπει να αποδώσουν καρπούς για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό θα ωφελήσει την ανάκαμψη, την αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 10% αν υπάρξει αυτή η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. No, no translation. uh -huh. it's no translation at all. There is translation, but But it, it's on English. Can I start again in Swedish? Θα ξεκινήσω και πάλι στα σουηδικά. Αργά. Yes, but it's better for me to speak in, in Swedish. Προτιμώ να μιλήσω στα σουηδικά. Μιλάτε λοιπόν συχνά και σε διάφορε περιστάσει για τι διορθωτικέ μεταρρυθμίσει ω απαραίτητε προσθήκε τη νομισματική πολιτική. σω λοιπόν κάπω να έκανα λάθο αυτά που άκουσα, αλλά δεν ακούω να μιλάτε για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ω σημαντικό παράγοντα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αυτό. Και αυτό μου προκαλεί έκπληξη, γιατί οι καλές μεταρρυθμίσεις για την ε, βελτίωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τις, ε, την ευρωπαϊκή οικονομία. Μία μελέτη καταδεικνύει ότι η ισότητα είναι καλή για την ανάπτυξη, για την αύξηση του ΑΕΠ σε ορισμένες περιπτώσεις σε επίπεδα μέχρι και 10%. Και θα ήταν πάρα πολύ θετικό να μπορούμε να εγγυηθούμε την ισότητα. Αυτό θα ήταν καλό και για την αγορά εργασία, γιατί έτσι θα μπορούσαμε πραγματικά να ε, εξαντλήσουμε το πλήρες δυναμικό όλων των ανθρώπων. Ναι, ναι, πρέπει να κλείσετε σιγά σιγά κυρία Λούτφιξεν. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το θέμα της ισότητας και γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ γιατί δεν μιλάτε πιο πολύ για θέματα ισότητας όταν πρόκειται για θέματα ανάκαμψης, ανάπτυξης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρώπη. Ναι, ευχαριστώ. Έγινε μάλλον λάθο ε, στη σειρά. Ένα λεπτό κύριε Κίρτσο, ένα λεπτό Σα παρακαλώ. Μόνο μία ερώτηση για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ε, αναπόφευκτα είναι ελληνική η ερώτηση. Ε, ίδια Κύριε Ντράγκη, εγώ θεωρώ ότι παίζετε πολύ θετικό ρόλο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Νότο και ειδικά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσει μεταξύ τη ελληνική πλευρά και των θεσμών όλοι ξέρουμε δεν πηγαίνουν καλά. Επειδή λοιπόν είστε άνθρωπο με μεγάλη επιρροή και κύρο, τι σκέπτεστε να κάνετε στην τελευταία κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων. Γιατί είναι τρει-τέσσερι οι παράγοντε που μπορεί να διαμορφώσουν τι εξελίξει και να αποτρέψουν μια αρνητική κατάσταση. Ε, θα μπορούσατε για παράδειγμα ε, να προτείνετε στην ελληνική πλευρά να δώσει έμφαση σε δύο-τρία σημεία, ε, αν όχι ο ίδιος, μέσα από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα μπορούσατε να γίνετε κάπως πιο ευέλικτοι στην τελική φάση ε, σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί φοβούμαι, εγώ εντάξει κάνω κριτική στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση είμαι, αλλά μήπως πάθουμε έτσι μια μεγάλη ζημιά όλοι μαζί, δηλαδή προσπαθώντας να κλείσουμε την ελληνική τρύπα ε, ανοίξουμε μια μεγαλύτερη μαύρη τρύπα για άλλες χώρες της, ε, της Ευρωζώνης. Νομίζω η κυρία Φερέιρα το έθεσε με τον τρόπο της. Επομένως, τι θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Συμφωνώ απολύτως και πλήρως με σας. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οπουδήποτε υπάρχουν στόχοι ισότητας ε, των δύο φύλων, τότε και η συμμετοχή στην οικονομία και η απόδοση είναι μεγαλύτερη. Τούτου λεχθέντος. Είναι βέβαια από τα τυπικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συζητήσει το θέμα αυτό στα πλαίσια των οικονομικών πολιτικών και των συζητήσεων για τις οικονομικές πολιτικές. Και μάλιστα μου έχουν ψηλοποιεί κιόλα ότι δεν πρέπει να πολύ μιλάω και για διερχοτικές πολιτικές κτλ. Κοιτάξτε, εμείς βεβαίως το κάνουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί οποτεδήποτε ε, υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ε, κύρια, στο κύριο μέλημά μα που είναι η σταθερότητα των τιμών, οπωσδήποτε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Παρεπιπτόντω, μπορώ να σα δώσω και πολλά παραδείγματα όπου τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 κεντρικέ τράπεζε αναφέρθηκαν ε, και μίλησαν ε, και αντιμετώπισαν ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην 2005. εντολή Ωστόσο, να σας πω και το εξής. Ο κανονισμός για την ε, ε, νομισματική οικονομική σταθερότητα ε, σε ορισμέ, μέσα από ορισμένε δικαστικές αποφάσεις στην ουσία διαλύθηκε. Βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα συμβεί το ίδιο υπό την αρμοδιότητα των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, δεν θα ήταν λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις ε, οι κεντρικές κυβερνήσεις ε, να είχαν ε, ορθώσει το ανάστημά τους κατά κάποιο τρόπο και να είχαν πάρει θέση έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτή η αρνητική επίπτωση. Αυτό νομίζω πρέπει να το έχουμε κατά νου ε, όταν ε, ε, αποφασίζουμε ποιες είναι οι διορθωτικές αλλαγές οι οποίες χρειάζονται έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερο δυναμικό ή καλύτερα αποτέλεσματα οικονομικά μια χώρα. Όσον αφορά την άλλη ερώτηση, δεν μπορώ να μπω στα λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές στην ουσία τώρα ε, θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να ε, φτάσουν σε μια ισχυρή συμφωνία η οποία μπορεί ε, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι να οδηγήσει σε συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα με κοινωνική δικαιοσύνη και με φορολογική βιωσιμότητα. Όπως είπα και στον ε, κύριο Φων Φάιτζάκερ προηγουμένως στην απάντηση που του έδωσα, υπάρχουν ε, ε, κάποια στοιχεία. Ένα το οποίο αφορά ας πούμε την τεχνική συμφωνία που είναι στην ουσία η ουσία του, του, της πολιτικής συμφωνίας και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αφορά την οικονομική συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ για την ανοιχτή σας διάθεση να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Πρέπει να πω ε, ε, επίσης ότι συμφωνώ με τα ε, ζητήματα τα οποία αναφέρατε και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τα σοφά σας λόγια. Ευχαριστώ. Dear colleagues, let's continue our meeting. I have some... Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μα, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω κάποιε ανακοινώσει να σα κάνω. Θα δώσω το, την Προεδρία στον πρώτο αντιπρόεδρό μα. Καταρχά, σε ό,τι αφορά τι συστάσει και τι αποφάσει που ελήφθησαν στη συνεδρίαση των συντονιστών στι 11 Ιουνίου να σας πω ότι ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ και ο Επιτροπός Μοσκοβίση θα παρουσιάσουν το πακέτο της Επιτροπής για την δημοσιονομική διαφάνεια σε κοινή ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Οίκων και Εντάξει, στις 2 Ιουλίου ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης θα προσκληθεί μαζί με τον Επιτροπό Μοσκοβισή για έναν ε, διαρθρωμένο διάλογο στις αρχές του Νοέμβρη και οι συντονιστές αποφάσισαν να προσκαλέσουν τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών προκειμένου να συναντηθούμε και να κάνουμε μια απόπειρα συμφωνίας επί ενός κειμένου το οποίο θα συγκεντρώσει μεγαλύτερη πλειοψηφία της Επιτροπής και στη συνέχεια να αναφέρουμε στους συντονιστές το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Συνάντηση του εισηγητή και των σκιωδών θα διοργανωθεί και οι σκιώδες όπως διευκρίνησα θα προσκληθούν επίσης. Η εικόνα θα προετοιμάσει η γνωμοδότηση για την έκθεση είναι για μία κοινή πράξη ε, ενωμένης ε, ψηφιακής αγοράς ε, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Στολογιάν θα παρευρεθεί στη Ρήγα στις 25 Ιουνίου και σε μία ημερίδα για το RFS 9. Επίσης συμφωνήσαμε να καλέσουμε εμπειρογνώμονες σε μία ακρόαση. Θα αποφασιστεί στο μέλλον η σύσταση της ακρόασης. θα βρείτε μία λίστα για τα ψηφίσματα που προτείνονται στα πρακτικά. Τέλος, μία ενημέρωση σε σχέση με τους τριμερείς διαλόγους. Καταρχάς, πολύ καλές ειδήσει έχουμε να αναφέρουμε γιατί ολοκληρώσαμε θετικά τον τριμερή διάλογο με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για τον κανονισμό για το ΕΦΣΥ. Θα το ψηφίσουμε αυτή την εβδομάδα από ό,τι ξέρετε και νομίζω ότι πραγματικά αποτέλεσε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στενό το χρονοδιάγραμμα επί το οποίο συμφωνήσαμε και θα βελτιωθεί σημαντικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη σε μεγάλο βαθμό την έντολη της, ε, των δύο επιτροπών για την οδηγία για την τριμερή διάλογο για την οδηγία για την διαμεσολάβηση για τις ασφάλειες. 8 Ιουνίου έγινε ο τριμερής διάλογος. Συμφωνήσαμε για το εύρος εφαρμογής της οδηγίας κατανολογία 200 όσο σε ό,τι αφορά τα, της επαγγελματική κατάρταξη, το έγγραφο ε, πληροφορίας προϊόντων για το χρονοδιάγραμμα και η επόμενη συνάντηση στα πλαίσια του διαλόγους διαλόγου στις 24 Ιουνίου για τις ε, Το Security Finance ε, ε, στον τρομερή διάλογο πετύχαμε σημαντική επιτυχία σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα στις 17 Ιουνίου επόμενη τριμερή διάλογος και τέλος ένας πρώτος διάλογος έγινε στις 2 Ιουνίου για τον κανονισμό για τα benchmark. Έγινε μια πρώτη αρχική συζήτηση στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και η Προεδρία θα καταρτήσει non-papers για τους συμβιβασμούς και προγραμματίζονται στις 15 Ιουλίου ε, περαιτέρω τριμερείς διάλογοι. Και τώρα θα δώσω το, την Προεδρία στον Μάρκο Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με το 4 της ημερήσια διάταξης. Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο Σβεν Γκίγκολτ είναι ο εισηγητής μας. Του δίνουμε τα χαρά στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα στραφώ στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να μοιραστώ μαζί σας την ε, απογοήτευσή μου γιατί τα μέσα ενημέρωση δεν ενδιαφέρουν για αυτή την τόσο σημαντική στατιστική έρευνα και έχουν φύγει. Αυτό είναι μια τεράστια παρεξήγηση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Επιτροπή μας. Αλλά, σε πάση περιπτώσει, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους κοιόδης εισηγητές, όλων των ομάδων που έχουν συμβάλει ενεργά, ο κύριος Τόρβαλτς, κύριε Γκάλπελτς, κυρία Μόσκα από τους σοσιαλιστές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό αντί να εστιάσω στις μεμονωμένες τροπολογίες να σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είχαμε μια συνάντηση των σκιωδών την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και μπορέσαμε να συμφωνήσουμε μεταξύ των παρόντων για ένα ενοποιημένο κείμενο και επίσης επειδή εδώ τίθενται πολύ τεχνικά εν μέρη προβλήματα, αποφασίσαμε να μεταθέσουμε σε την ψηφοφορία κατά μία εβδομάδα και επομένω έχω ζητήσει να μην ψηφίσουμε αύριο, ώστε οι ομάδες εργασία των διαφόρων πολιτικών ομάδων να έχουν τον χρόνο να συζητήσουν τι συμβαστικέ λύσει των σκιωδών εισηγητών αυτό δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω γραφειοκρατία βέβαια, γιατί μάθαμε από την Λετωνική Προεδρία ότι το θέμα αυτό δεν θα μπορέσει να περατωθεί μέσα στη Λετωνική Προεδρία, αλλά μόνο στην επόμενη. Δεν χάσαμε λοιπόν, δεν χάνουμε τίποτα με το να μεταθέσουμε κατά μία εβδομάδα το θέμα αυτό επί της ουσίας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά τους και τη γενική υποστήριξη που έχουν δώσει με τις προτάσεις τους σε όλα τα θέματα ουσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των στατιστικών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θεσμών αυτών σε ορισμένα θέματα διακυβέρνησης για τα στατιστικά συστήματα. Η κύρια συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών η οποία φαίνεται και από τις τροπολογίες, έχει εστιάσει στο θέμα του εφικτού να υπάρξουν βελτιώσεις ως προς το άρθρο 5 και πάλι επί τη βάση τροπολογιών του ΕΛΚ και των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έχουμε προχωρήσει σε μια συμβαστική λύση που λέει ουσιαστικά ότι οι στατιστικές βελτιώσεις θα οδηγήσουν σε πιο λεπτό, λεπτόκοχη κατά κάποιο τρόπο ανάλυση των στοιχείων σε σχέση με τους ε, πραγματικούς δικαιούχους των ε, χρηματοπιστωτικών φορέων και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις και να εισαχθεί η δυνατότητα για την Κομισιόν να υπάρξει δυνατότητα αυτοεξέλισης, opt-out, εάν δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση για να γίνει αυτό αποτελεσματικά. Και επίσης στην ε, πιλωτική μελέτη θα πρέπει να εξεταστεί όχι μονάχα η μεθοδολογία που θα πρέπει να δοκιμαστεί, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η συγκρισιμότητα και το λογικό κόστος και το εφικτό αυτών των αλλαγών. Πέραν αυτού, έχουμε συμπεριλάβει και μια τροπολογία των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και επίσης στις συμβαστικές ε, <clears throat> τροπολογίες έχουμε κάποιες τροπολογίες που κάνουν σαφές, μία από τους φιλελεύθερους συγκεκριμένα, ότι δεν θα πρέπει να προκύψει υπερβολικό και περιττό άχθος και πρόσθετο στατιστικό άχθος πέραν αυτών που έχουν να κάνουν με τα απολύτως απαραίτητα. Συμπεριλαμβάνω επίσης και μια πρόταση από τους φιλελεύθερους και από άλλες ομάδες μια αλλαγή που δίνει τρία, τρεις μήνες για τον έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων και την συνήθη φρασιολογία ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ότι η καταξιοδότηση πράξη έρχονται στο Κοινοβούλιο λίγο πριν από τις διακοπές, κάτι το οποίο μειώνει τον ουσιαστικό χρόνο ελέγχου. Και επίσης στη συμβαστική θέση έχουμε συμπεριλάβει εκφράσεις από τους πράσινους και τους συντηρητικούς για να χρησιμοποιηθούν οι τελευταίες καινοτομίες, ιδίως σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για τα στατιστικά συστήματα. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο δεν έχουμε ακόμα επιλύσει πλήρως αφορούσε μια τροπολογία των σοσιαλιστών που ζητούσε, για να το πω επίοικος, να υπάρξουν αντικίνητρα για τα κράτη-μέλη να παρουσιάζουν ωρεοποιημένα στατιστικά στοιχεία. Εγώ κατανοώ αυτή την τροπολογία και την υποστηρίζω, αλλά νομίζω ότι ποτέ τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν ποτέ σε επίπεδο συναπόφαση να συνενέσουν σε μια τέτοια ρήτρα Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να υπάρξει μια τέτοια διάταξη στην έκθεσή μας, απλώς μονάχα θα οδηγήσει σε μακροσκελείς διαμάχες και συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Όπως, όπως είπα λοιπόν, αν θέλει η σοσιαλιστική ομάδα να διατηρήσει αυτή την τροπολογία, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα που θα έχουμε με το Συμβούλιο και το γνωρίζουμε και από τις συζητήσεις με τη Eurostat ότι η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων δεν είναι πάντα ισόμορφα ε, υψηλή από όλα τα κράτη-μέλη. Επομένως το να μιλήσουμε για αντικίνητρα σε σχέση με τα κράτη-μέλη δεν είναι ίσως η πιο εύστοχη στάση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν συνεργαστεί μαζί μου για αυτή την τόσο συναρπαστική έκθεση και προσβλέπω στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε και να δώσουμε το λόγο στους Σκιώδης από το ΕΛΚ στην κυρία Γκαλπέλτς καταρχάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή με τον εισηγητή. Ήταν πραγματικά εξαιρετική και ήταν πολύ χρήσιμες οι τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση με τα στατιστικά στοιχεία να παρακολουθούμε τις αλλαγές. Όλα καλά, ρωτάει η ομιλήτρια με την ναι. Μάλιστα. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνονται μόνο αλλαγές που δεν θα προκαλούν μεγάλε διαφορετικέ τροποποίησεις. Και γι' αυτό λοιπόν καταθέσαμε κάποιες τροπολογίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τις αποδέχτηκε ο εισηγητής. Συγκεκριμένα εδώ μιλάμε για τη συλλογή δεδομένων, μιλάμε για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και μιλάμε για έργα εξάντε, για πληθυκά τέτοια έργα Αν λοιπόν όντως τα έργα αυτά αποδειχτούν ότι είναι αποτελεσματικά, μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Ξέρουμε λοιπόν όλοι ότι το τελευταίο καιρό οι διεθνείς ε, ροής κεφαλαίων είναι πολύ περίπλοκες και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσουμε. Μας βοηθούν λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία εκείνα όπου είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία τους. Άρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην διάσταση της ποιότητας. Οι τροπολογίες είναι όντως πολύ θετικές. Ε, δύο μόνο είναι ίσως αφιλεγόμενες. Και εδώ δεν είναι τέλειο το αποτέλεσμα θα έλεγα. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το άρθρο 20 για το απόρριτο, confidentiality. Ε, εδώ το ECR κατέθεσε μια πρόταση η οποία θεωρούμε ότι είναι καλή. Σε ό,τι αφορά τα πέναλτις της κυρώσης. Τα αντικίνητρα, disincentives, τα οποία ανέφερε και ο εισηγητής. Πιστεύω ότι είναι καλά και χρήσιμα, αλλά συμφωνώ και με τον εισηγητή ότι δεν θα τα αποδέχονταν τα κράτη-μέλη. Και στο σύνολό τους πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τις συμβαστικέ λύσεις και θα τις υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κ. Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αλέσια Μόσκα δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ στην Επιτροπή και μου ζήτησε ε, να, να σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις ε, των σοσιαλιστών για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για την εργασία του, καθώς επίσης και όλους τους σκιώδεις για αυτή τη διαδικασία που ελπίζουμε ότι θα τελειώσει με ένα συμβαστικό κείμενο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτόν τον κανονισμό να γίνει νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε ε, οι στατιστικές να είναι διαφανείς, ε, καλύτερες και επομένως ε, να βελτιωθεί το σύνολο της οικονομικής πολιτικής και η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί με την ανάγκη αυτές οι στατιστικές, κυρίως δε οι ροές κεφαλαίων, να αναφέρονται σε ακαθάριστες ροές και σε καθαρά ε, ποσά τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιες είναι οι ροές ε, των κεφαλαίων με τρόπο ώστε ε, να καταπολεμάται η φοροδιαφυγή. Η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος δημοσίευσης αυτών των στοιχείων ε, έτσι ώστε να παρακολουθούνται από κοντά οι ε, στατιστικές σε συνεργασία ε, και με τα όσα γίνονται στον ΟΣΑ, στο Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο ή και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Επίση, η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της ε, Eurostat και ε, το σύνολο των ε, οικονομικών φορέων και βεβαίω και οι σχέσεις με τις, ευρωπαϊκές, με τις κεντρικές τράπεζες έτσι ώστε οι στατιστικές να αναλύονται με καλύτερο τρόπο. Επίσης, η σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί να δοθεί η δυνατότητα στην Κομισιόν Λοιπόν να προετοιμάζει κατεξουσιοδότηση πράξη, έτσι ώστε να, οι στατιστικές να είναι καλύτερες. Τέλο, η συνέλεφο Μόσκα αλλά και ε, το σύνολο της ομάδας ε, είναι αρκετά ικανοποιημένο από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία και να σας πω ε, και εγώ ότι η τροπολογία σχετικά με την δυνατότητα επιβολή κυρώσεων σε χώρε διότι δεν, δεν ενεργούν σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό. Είναι ένα ζήτημα, λέω, αυτών των κυρώσεων που θα πρέπει ε, να συζητήσουμε και σε, σε μελλοντικές ε, συνεδριάσεις. Αλλά ε, θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι και η θέση της, του Συμβουλίου, όπως σύμφωνα και με αυτά που είπε και ο συνάδελφος Γκίγκολ στην αρχή της παρέμβασής του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες απαιτήσει του Συμβουλίου, του συγγνώμη, του Κοινοβουλίου ίσως θα είναι πιο εύκολο να ληφθούν υπόψη και είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει τα μέτρα αυτά τα οποία θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απαιτήσει, οι οποίες μοναδικό στόχο έχουν τη βελτίωση της διαφάνειας και της σοβαρότητας των στατιστικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ECR. Κανείς? Δεν είναι εδώ ο κ. Καμάλ. Για τους φιλελεύθερους, ο κ. Τόρβαλτ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ακολουθήσω τον εισηγητή. Μιας και αυτός μίλησε αγγλικά. Γιατί θα ήταν δύσκολο να τα πω όλα αυτά στα γερμανικά. Μα εξαιρετικά τα λέτε στα γερμανικά. Όπως και να έχει. Όπως είπε και ο Σβέν στην παρουσίαση του, όπως ακούσατε, ήταν εξαιρετικός ως ο εισηγητής. Κατάφερε να πετύχει το κατόρθωτο σε κάποιες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Ευχολόγιο. Χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο στα γερμανικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γίγκολτ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Τόρματς, λέει ο πρόεδρος, για την ΚΟΕ. Βίγκας. Ευχαριστώ πολύ. Μια πρώτη τεχνική παρατήρηση φυσικά συμφωνούμε σε όλες τις τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των στατιστικών που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, τον Ευρωστάτ μαζί με τους Εθνικούς Στατιστικούς Οργανισμούς. και γι' αυτό υποδεχόμαστε θετικά πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του κ. Γκίνγκολτ. Τονίζουμε ιδιαίτερα τη σημασία του να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αντικατασταθεί η Επιτροπή για, την, για, την, ε, για το ισοζύγιο πληρωμών από την Επιτροπή Στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε επίσης να βελτιωθεί η ε, ποιότητα των δεδομένων σε σχέση με τις ροές κεφαλαίων, ξεχωρίζοντας τις ροές οι οποίες αφορούν τη δημιουργία πάγιου κεφαλαίου, δηλαδή των επενδύσεων, των πραγματικών επενδύσεων, από τα κεφάλαια τα οποία είναι απλώς κινήσεις κεφαλαίων και τίποτα παραπέρα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το σύστημα να παρακολουθεί και όλα τα επίπεδα καταπολέμησης της ε, απάτης και του ξεπλήματος χρημάτων, γιατί έχουμε εδώ πέρα μια πολυπληθώρα νέων κανονισμών που οδηγούν σε περισσότερα δεδομένα, τα οποία όμως παρόλα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη από το σύστημα. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό επίσης να περιορίσουμε να μην τροποποιείται σε ένα παράτημα η διάταξη αυτή για, τους, ε, για τις χρηματικές ροές, να μην με τη μέθοδο αυτή ουσιαστικά υποσκαφθεί αυτή, η, αυτό το νομοθέτημα και τώρα ένα πιο πολιτικό κομμάτι των παρατηρήσεών μας θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πρόταση αυτή γιατί μιλάμε για την πρόταση αλλαγής ενός κανονισμού που έχει κέριο χαρακτήρα <clears throat> και που παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική διακυβέρνηση και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτός ο μηχανισμός να εξακολουθεί να λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι άδικος, είναι πηγή πολλών από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες μας, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η οικονομική διακυβέρνηση, τίγει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την οικονομική ευρωστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Άλλοι συναδελφοί, δεν ζήτησε κανείς άλλο το λόγο. Θέλει κανείς από την Επιτροπή το λόγο από τη γυροστάτ, ή από την ε, Κεντρική Τράπεζα. Thank you. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα με χαρά να σας ανακοινώσω ότι είμαστε ικανοποιημένοι που η πρόταση της Επιτροπής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία τα απαραίτητα και χαρακτηρίζεται από επικοδομητικές συζητήσεις. Είπαμε εξ αρχής ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ευελιξία για να διορθώνονται ε, οι απαιτήσει σε ό,τι αφορά τα δεδομένα σε δίθεση επίπεδο. Και διάφορες από τις τροπολογίες ε, που προτάθηκαν προβλέπουν άλλες δυνατότητες για το άρθρο για τις πράξεις κατεξουσιοδότησης εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης του κειμένου προκειμένου να εξυπηρετούνται τα διάφορα συμφέροντα των θεσμών. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες τροπολογίες για το FDI. Με μεγάλο ενδιαφέρον τις κοιτάμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξετάσουμε την δυνατότητα έχουν γίνει κάποιες μελέτες ε, για τα θέματα αυτά. Και θα μπορούσαμε να τις συνεχίσουμε για να πετύχουμε την εφαρμογή. Θα ήθελα να θέσω το θέμα της ενδεχόμενης επιβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων για τα στατιστικά στοιχεία. Η πρόταση όσο έχει τώρα, αυτή τη στιγμή, θέτει προηγούμενο. Γιατί στην παρούσα φάση υπάρχει μόνο μία διάταξη που περιλαμβάνεται στο six-pack για την οικονομική διακυβέρνηση. Στο άρθρο 8 του κανονισμού 1173 του 2011 που δίνει άμεσο δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει κύρωση σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει σκόπιμη παρερμηνία ή σοβαρή αμέλεια στατιστικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις αυτό, αυτές δεν ε, ισχύουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, όπως προβλέπονται από τις συνθήκες. Υπάρχει και μια άλλη διάταξη ωστόσο στον κανονισμό 223 που εγκρίθηκε προσφάτως στο άρθρο 12 παράγραφο 5 που δίνει εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει ενδεχόμενες υποθέσεις παραποίηση στατιστικών δεδομένων. Και στη συνέχεια ασφαλώς να προβεί σε τεκμεριωμένη έκθεση προς το Συμβούλιο με την τελική απόφαση κατά πόσον χρειάζονται ή όχι κυρώσεις. Να επιστήσουμε την προσοχή σας λοιπόν στη δυνατότητα αυτή που προβλέπετε στον κανονισμό 223 αποτελεί και αυτό έναν τρόπο να πετύχουμε ενδεχομένω τον ίδιο στόχο. <coughs> Τέλος, δε. Προσβλέπουμε την έναρξη, την των ε, τριμερών διαλόγων με την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου ενδεχομένω. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους ε, για τα ευγενικά τους λόγια. Ε, εν συντομία να, ξαναδούμε τα ζητήματα ε, τα οποία σχετίζονται με, την, με το άρθρο 20 και το, ε, το σεβασμό του απορρίτου και της εμπιστευτικότητας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας διαφοροποιεί. όσον αφορά το, τα όσα είπε ο κύριος Φερνάντες, και οι σοσιαλιστές σχετικά με τις κυρώσεις. Ε, το ανέφερε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγο. Όπως είπα και προηγουμένως, έστω και αν ε, υπάρχει μονάχα ένα τέτοιο προηγούμενο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εγείρει τέτοια αξίωση. Πρέπει να πω ότι με αρκετό ενδιαφέρον βλέπω το ζήτημα αυτό από όταν ξεκίνησα ως εισηγητής προπολογισμού για την Επιτροπή μας, γιατί εκεί διαπίστωσα ότι για να καλυφθούν οι στατιστικές δεσμεύσεις ε, ε, υπάρχουν ε, νόμοι νόμοι ε, που ε, ανταποκρίνονται σε προηγούμενες αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να στηρίξω αυτό που λέτε, να το υποστηρίξω έστω και αν πιστεύω ότι ε, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουμε πολιτικά και νομικά προσκόμματα. Απάντως είναι ένας ενδιαφέρον διάλογος όσον αφορά την αναφορά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Νίλδης. Ε, τα Χριστούγεννα είναι πολύ σημαντικά, ωστόσο πιστεύω ότι ε, ε, ε, πραγματικά πέρα και εγώ με σκεπτικισμό βλέπω το ενδεχόμενο ε, να απολούνται χριστουγεννιάτικα προϊόντα εκτός χριστουγεν, χριστουγεννιάτικης περίοδου και εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω τελειώνοντας ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κάνουν διάφοροι συνάδελφοι βασίζονται σε υφιστάμενη εργασία, βασίζονται σε πράγματα τα οποία έχει δώσει δώσει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, οι φυστάμενες ε, μελέτες κλπ. Ε, εν μέρη εργασίες και μελέτες που έχει κάνει το Διεθνές Ταμείο και αυτό που θέλουμε είναι τώρα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να επιταχύνουμε την υλοποίηση θεμάτων τα οποία έχουμε ήδη επεξεργαστεί. Από ό,τι είδα δεν έχετε υποβάλει τροπολογίες και επομένως ε, θεωρώ ότι στηρίζετε αυτά που κάνουμε. Τέλος, ε, όσον αφορά την Κομισιόνου και τα όσα είπε σχετικά με την απαραίτητη ευελιξία. Πρέπει να επιμείνω ότι το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα δεν έχει ε, πει ότι θέλει να περιορίσει σε οποιοδήποτε βαθμό την ε, ευελιξία. Δεν συμφωνούμε λοιπόν ότι γίνονται σημαντικές τροποποιήσεις ε, χωρίς, την δυνατότητα, ε, χωρίς να έχει δυνατότητα ο συνομοθέτης να δει τις αλλαγές αυτές. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Το Κοινοβούλιο δεν θα παρέμβει εάν όλα πάνε καλά. Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη ευελιξίας, εμείς αμφισβητούμε, θέτουμε ένα αμφιβόλα κατά κάποιο τρόπο και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Θέτουμε σε αμφισβήτηση λοιπόν το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι της ε, νομοθεσίας γίνεται de facto και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να μπορεί ο συνομοθέτης να εκφράσει την άποψή του και στις αυριανές συζητήσεις ε, νομίζω ότι θα το ξανασυζητήσουμε αυτό, αυτές τις δηλαδή de facto ε, αποφάσεις οι οποίες αποκλείουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ και οπωσδήποτε θα δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό και σε πολλούς συναδέλφους και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ Σβέν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα στον τριγωνικό διάλογο. Έχουμε εμπειρία από άλλα θέματα γι' αυτό. Η, έχει εκπνεύσει η ψηφοφορία θα γίνει σε 10 μέρες με την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή μας. Ερχόμαστε κατευθείαν στο σημείο 5 της ημέρας της διάταξης που είναι το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Δομών και Επενδύσεων και τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το άρθρο 23 της εφαρμογής των κοινών κανόνων με εισηγητή τον κύριο Κίρτσο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω πάρει πολύ ενδιαφέρουσε τροπολογίε από του συναδέλφου μα σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότηση που θα δώσουμε ως Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων στην Επιτροπή ΡΕΤΖΙ, την Περιφερειακή Επιτροπή, σε σχέση με, το ευρωπαϊκό, με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Διάρθρωσης και Επενδύσεων. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις κατευθυντήρες γραμμέ για την εφαρμογή του άρθρου 23 των κοινών κανόνων. Του αρμόδιου κανονισμού οι περισσότερες τροπολογίες έρχονται από δύο διαφορετικές πολιτικές θεωρίες. Υπάρχουν αυτοί και περιλαμβάνω και τον εαυτό μου σε, στη μία άποψη που πιστεύουν ότι χρειάζεται μια υγιής μακροοικονομική και δημοσιονομική πολιτική και η ενίσχυση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρησιμοποιηθούν πλήρω <clears throat> οι ευκαιρίε που δημιουργούνται από τα ταμεία επενδύσεων και διαδοτικού χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δίνουν περισσότερη έμφαση στις κοινωνικές και περιφερειακές πτυχές. Ζήτησα να γίνει μια συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για να βρούμε ενδεχόμενα τροπολογίες συμβασμού, γιατί έχουμε 62 τροπολογίες για τις 5 παραγράφους. Είναι φανερό ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή γλώσσα, χωρίς να δημιουργήσουμε σύγχυση για τους στόχους που επιδιώκουμε. Δυστυχώς οι σκιώδεις εισηγητές δεν μπορούσαν να συναντηθούν όταν το είχα προτείνει, την ημέρα που το έχω προτείνει. Γι' αυτό θα κάνω μια γραπτή ανταλλαγή απόψεων. Θα προσπαθήσω να διατυπώσω ένα σύνολο συμβαστικών τροπολογιών μέχρι την Πέμπτη και να τις διαβιβάσω σε όλους τους ενδιαφερομένους συναδέλφους, ώστε στην αρχή της επόμενης εβδομάδας να ξέρουμε πού μπορούμε να έχουμε μια κοινή διατύπωση και για ποιες παραγράφους θα πρέπει να διαβιβάσουμε φωνήσουμε και να ψηφίσουμε. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο κύριος... Ε, ο κύριος Γιώργος Φερνάντης Αλβάρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξαναμιλήσω κι εγώ για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής ομάδα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, καθώς επίσης ε, και τους ε, σκιώδες εισηγητές. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε να βρεθούμε έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις και να προχωρήσουμε το κείμενο. Πιστεύω ότι είναι επί ισορροπημένης βάσης η πρόταση του εισηγητού. Ωστόσο θα ήθελε η Σοσιαλιστική Ομάδα να επιμείνει επί δύο θεμάτων τα οποία συζητήσαμε συζητήσαμε ε, και σε ανταλλαγή απόψεων πριν από τούτη τη συζήτηση. Το πρώτο ο καθορισμός ε, σαφών ορίων ε, όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 23 ε, σε σχέση με περικοπές των διαδοτικών ταμείων σε χώρες. Χώρες οι οποίες δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της μακροαιρεσιμότητας. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να γίνεται η σωστή αξιολόγηση ε, να, ε, ξεκινώντας από υπερβολικό έλλειμμα μέχρι να φτάσουμε στις ε, κυρώσεις. Δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα διευθυντικά ταμεία έτσι ώστε να κυρωθούν ακόμα περισσότερο οι χώρες οι οποίες ήδη δεν καλύπτουν κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως. Όλα αυτά προβλέπονται και στο, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά εμείς θέλουμε ένα κείμενο στο οποίο η δυνατότητα προσφυγής και χρήσης του άρθρου 23 να είναι περιορισμένη. Το δεύτερο το οποίο ενδιαφέρει την πολιτική μου ομάδα είναι να καθοριστεί σαφής ε, ε, διαδικασία σε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 23. Σε αυτή την περίπτωση να χρειάζεται η διαβούλευση και η συμμετοχή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και ε, σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείται το άρθρο 23 σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για την οικονομική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προτείνουμε βεβαίως συμβιβαστικό κείμενο και τέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή αλλά και όλους τους σκιώδεις για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο Στάνισλαφ έχει το λόγο για το ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχοντας διαβάσει τις τροπολογίες, μπορώ να δω ότι οι περισσότερες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Επομένως, συμπεραίνω ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά τον ρόλο των διαφθορτικών ταμείων και των διαφθορτικών πολιτικών τους βασικούς στόχους και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των ταμείων. Αντίθετα από τον εισηγητή, εγώ εκπροσωπώ μια διαφορετική άποψη σε σχέση με τον ρόλο σε σχέση με το επίπεδο της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εθνικών κρατών για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Αυτό οφείλεται στην προηγούμενη μου καριέρα γιατί ήμουν επικεφαλής τοπικής αυτοδιοίκησης και για πολλά χρόνια. Επίσης <clears throat> ήμουν υπεύθυνο σε περιφερειακό επίπεδο. Οι περισσότερες τροπολογίες τονίζουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση να δοθεί στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Κάποιες τροπολογίες ορθώς, κατά την απόψή μου, τονίζουν ότι ο τελικός δικαιούχος των διαρθωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι οι πολίτες οι τοπικέ κοινότητε. και όχι τα κράτη-μέλη. Αυτά καθε αυτά. Για αυτό το λόγο, το να επιτύχουμε το στόχο της πολιτικής συνοχής δεν έχει να κάνει μονάχα με την ικανότητα μια κεντρική κυβέρνηση να εκπληρώσει τους στόχου της σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συνάδει με την ικανότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων που απαιτούν οι διάφορες περιφέρειες και περιοχές. Φοβάμαι ότι αν αναπρογραμματίσετε τις δραστηριότητες αυτές θα υπάρξει χειρότερη κατάσταση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό υποστηρίζω όλες αυτές τις τροπολογίες οι οποίες ορθά <clears throat> υπογραμμίζουν ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια πλήρη αξιολόγηση και δικαιολόγηση εάν υπάρχει επαναπρογραμματισμός και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αποτελεσματικότητας σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν και την αρχή της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η έλλειψη χρηματοδότησης θα οδηγήσει σε σώρευση περισσότερων προβλημάτων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. <clears throat> Συγχρόνως όμως να υπογραμμίσω ότι παρά το γεγονός ότι συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει μια κατάσταση όπου οι τοπικές αρχές φέρουν αυτομάτως το βάρος των αποφάσεων που λαμβάνονται στο εθνικό επίπεδο, δεν μπορώ να υποστηρίξω και τις τροπολογίες οι οποίες διαγράφουν οποιαδήποτε έννοια σωστής διαχείρισης, γιατί η σωστή οικονομική διαχείριση είναι μία από τις προϋποθέσεις για μία πολιτική συνοχής που λειτουργεί σωστά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε περιπτώσεις όπου οι τελικοί αποδέκτες των κονδυλίων, οι περιφέρειες, οι κύριοι πολίτες χάνουν αυτή τη χρηματοδότηση που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη σχεδίων και την οικονομική ανάπτυξη περιφερειών και κοινοτήτων. Βέβαια, τα κάτι μελη είναι υπεύθυνα για να εξασφαλίσουν τη σωστή διαχείριση των οικονομιών τους. Και όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, εγώ υποστηρίζω τις τροπολογίες οι οποίες θα ενισχύσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους φιλελεύθερους δεν βλέπω το σκιώδη εδώ. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Από την ΚΟΥΗ, ο κύριος Παπαδημούλης. Θα πάρτε το λόγο όμως εσείς, Μαρίζα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες που τις γνώριζε βέβαια ο και ξέρει και ποια είναι η θέση μας που δεν συμφωνεί με την αρχή που έχει διατυπώσει ο ίδιος για την εφαρμογή του άρθρου 23 σε σχέση με τους κοινούς κανόνες η δική μας άποψη είναι ότι η χρήση του άρθρου 23 για να περικοπούν τα διαφορετικά ταμεία προς τις χώρες οι οποίες ε, καθορίζονται από κριτήρια άλλων νομοθετικών μέτρων, αυτό είναι μια διπλή κύρωση στις χώρες αυτές, γιατί μιλάμε για χώρες οι οποίες χρειάζονται τα διαφορετικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής, αλλά οι χώρες αυτές ήδη έχουν υποστεί πρόστιμο μέχρι και 2% του ΑΕΠ για το γεγονός ότι δεν έχουν ικανοποιήσει τα κριτήρια αυτά που αναφέραμε. Αυτό απλώς θα επιδεινώσει την κατάσταση ανισότητας και ανισομέρειας μεταξύ των διαφόρων οικονομιών της ε, ζώνης της, ε, του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι μια βαθιά αντίφαση και γι' αυτό δεν δεχόμαστε μια τέτοια προσέγγιση δεν δεχόμαστε λοιπόν καταρχήν αυτήν την αρχή της μακροερεσιμότητας, αλλά περαιτέρω αυτού το να συνδέσουμε την αρχή της μακροοικονομικής ερεσιμότητας στην πολιτική διαρθρωτικών πόρων και συγχρόνως στο σύμφωνο ανάπτυξης και σταθερότητας, αυτό είναι ακριβώς μια κατάσταση που μας οδηγεί στο χειρότερο όλων των δυνατών κόσμο. Γιατί ο στόχος της πολιτικής συνοχής, ο στόχος των διαφθορτικών πόρων δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι να επιβληθούν προϋποθέσεις ή οικονομικές κυρώσεις μακροοικονομικού χαρακτήρα που προφανώς θα έχουν σε συνέπεια να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένε περιφέρειες και θα θίξει κράτη-μέλη και περιφέρειες που ήδη έχουν ξεκινήσει σε ένα μειονεκτικό επίπεδο. Αυτό που πρέπει να κάνει το Ταμείο Συνοχή είναι ακριβώ το αντίθετο. Να ακολουθήσει αυτή τη βασική αρχή του να εξασφαλίσει, να επιδιώξει μια ισορροπημένη ανάπτυξη η οποία θα μειώσει τι ανισότητε όταν υπάρξει πραγματική σύγκριση μεταξύ χωρών και περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε ένα μηχανισμό ο οποίο θα επιδεινώσει τι ε, διαφορέ αυτέ αντί να επιτύχει την πραγματική σύγκριση Γι' αυτό το λόγο η θέση μας <clears throat> είναι ότι θα πρέπει να αναστα... ότι η αναστολή των χρηματοδοτήσεων προς τα κάτι μελη που βρίσκονται σε δυσκολίες θα έχει σαν μόνο αποτέλεσμα να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο αυτές τις δυσκολίες που διατρέχουν. Ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε απόφαση η οποία έχει να κάνει με αναστολή πληρωμών για τα διαφορετικά ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να λαμβάνεται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος, ότι τα ποσά δεν χρησιμοποιούνται για τα σωστά ε, σχέδια, ότι υπάρχουν ατασταλίες ή μη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων σε καμία όμω περίπτωση δεν θα πρέπει να συνάπτεται με την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ένα κράτος μέλος. Για μένα αυτό είναι ένα κεφαλαιόδες θέμα και εδώ <clears throat> βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες ε, αντιφάσεις που υπάρχουν στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται μόνο προς την ε, πειθαρχία και τις κυρώσεις για τους ε, πιο αδύναμους, αλλά δεν κάνει τίποτα για να επιλύσει τα προβλήματα των ανισοτήτων ή τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι πιο ασθενείς οικονομικές, ε, οικονομικά χώρες, που για μας πρέπει να είναι αυτός ο στόχος των ε, πολιτικών συνοχής και διαφορετικών και όχι η επιβολή κυρώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους πράσινους, ο Σβεν Γκίγκολτ δεν είναι παρόν και έτσι περνάμε στην ομάδα του EFTD. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφου Βάλλη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Ε, αλλά θα μεταφέρω τα κύρια σημεία επί των οποίων ε, βασίζεται η θέση της πολιτικής μας ομάδας. Θα επανέλθω σε αυτό που έλεγε πριν η συνάδελφος ξεκινώντας από μια βασική αρχή που κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι ε, σαφή στα πλαίσια του της έκθεσης. Με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η στάση πληρωμών ε, του Ταμείου Συνοχής σε περίπτωση, παρά σε περίπτωση απάτης, διαφθοράς ε, ή παρίσφρησης του οργανωμένου εγκλήματος στη διαχείριση ε, των χρημάτων αυτών. Αυτές ε, είναι οι περιπτώσεις τις οποίες ε, μπορεί να σταματήσει η καταβολή των χρημάτων από το Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει να είναι σαφές αυτό. Επίσης, σαφής θα πρέπει να είναι ο στόχος των πόρων του Ταμείου Συνοχής, που δεν είναι άλλος από την προσέγγιση των δικών περιοχών της Ευρώπης προς τις πιο πλούσιες περιοχές της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι αν εφαρμόσουμε το άρθρο 23 του κανονισμού, όχι μονάχα δεν θα επιτρέψουμε αυτή την προσέγγιση, δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν ε, την επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά αντιθέτως ε, θα δυσχεράνουμε έτσι περαιτέρω την κατάσταση. Ε, η ερεσιμότητα τώρα, σε σχέση δηλαδή με τους κανόνες μακροοικονομικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι ο συσχετισμός με το, κανόνα, με το άρθρο 23 δεν είναι σωστός. Ε, μία χώρα η οποία δεν ε, ε, μπορεί να καλύψει κάποιες προϋποθέσεις ήδη υφίσταται κυρώσεις. Επίσης στο άρθρο 23 υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα κατά την άποψή μας. Αυτό το άρθρο βασίζεται σε αξίες ας πούμε όπως το ΑΕΠ μιας χώρας. Είναι όμως σαφές ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους γίνεται κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή του κεντρικού κράτους. Έχουμε, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε περιπτώσεις όπου ε, η, το ΑΕΠ και η τρύπα του ΑΕΠ να έχει προέλθει από τη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά οι επιπτώσεις ε, του άρθρου 23 ε, να αφορούν τις περιφέρειες, οι οποίες όμως είχαν χρηστή διαχείριση. Υπάρχει ακόμα και άλλο ένα σημείο, το τελευταίο, το οποίο ε, θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια ε, αυτής, ε, αυτού του κειμένου. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη μας από ό,τι φαίνεται το αίτημα επαναπρογραμματισμού των συμβάσεων οδηγεί σε σημαντικά διοικητικά έξοδα τα οποία τελικά αφορούν τις περιφέρειες και τους τοπικούς οργανισμούς. Άρα επιπλέον επιβάρυνση αυτών των οργανισμών. Ε, θα ήθελα να ζητήσω να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, σοβαρά ε, λάθη τα οποία έχουμε ήδη κάνει στην αντιμετώπιση των χωρών οι οποίες ακόμα τώρα ε, προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χώρες οι οποίες είναι σε ύφεση και σε λιτότητα ε, να επιβαρυνθούν διπλά μέσα από τέτοιου είδους ε, μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Υπάρχει κανένας που να θέλει να λάβει το λόγο ακόμα. Είναι μια γνωμοδότηση βέβαια που πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω η Κομισιόν αν ήθελε να λάβει το λόγο στον εισηγητή. Θέλετε να πείτε κάτι ή η η να πει κάτι Πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση, τον εισηγητή και τους διάφορους σκιώδεις εισηγητές. Ε, δύο-τρία δύο, σχόλια μονάχα. Πρώτα απ' όλα, η ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται στη λεγόμενη πρώτη πτυχή του άρθρου 23 της παραγράφους 1 έως 6 γιατί ακολουθεί τη δήλωση της Κομισιόν. Η ανακοίνωση αυτή όταν είχε, είχαν εγκριθεί, εγκριθεί ο κανονισμός για τους κοινού κανόνες και δεν αφορά το σύνολο του άρθρου 23, αφορά μονάχα τις έξι πρώτες παραγράφους του άρθρου 23. Δεύτερον, η Κομισιό θέλει να επαναλάβει ότι εμείς θα δώσουμε μεγαλύτερη σταθερότητα, θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα και δεν θέλουμε να έχουμε συχνό αναπρογραμματισμό για λόγους ότι καταρχήν πολλές φορές τα προγράμματα τα οποία υποβάλλονται θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αναχώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και επίσης θα θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρχει πρόσθετο διοικητικό κόστος λόγω του επαναπρογραμματισμού. Τρίτον, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα της ε, αναστολής των πληρωμών φυσικά θα λαμβάνονται υπόψη και η ανακοίνωση της Κομισιόν λέει ότι μια ενδεχόμενη αναστολή θα πρέπει να γίνεται με τρόπο αναλογικό και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο κράτος μέλος και επομένως θα πρέπει να εφαρμόσουν οι λεγόμενοι ε, παράγοντες μετριασμού που αναφέρονται στον κανονισμό αυτό σε περίπτωση αναστολής των ε, χρηματοδοτήσεων και επίσης θέλουμε να διατηρήσουμε τις ε, διαταραχές στο ελάχιστο για να μειώσουμε και το διοικητικό κόστος και τέλος θέλω να διευκρινίσω γιατί η ανακοίνωση δεν λέει τίποτα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού <clears throat> Κοινοβουλίου απλούστατα γιατί στη δήλωση που ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2013 η Κομισιόν όπου δεσμεύτηκε στο να εγκρίνει αυτήν την ε, ανακοίνωση ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιλαμβανόταν σε αυτήν την ανακοίνωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω στο λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Κίρτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι λίγο πολύ θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Χρειαζόμαστε όμως ε, μια επιταρχημένη και αποτελεσματική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε και μια κοινωνικά υπεύθυνη και κοινωνικά ευαίσθητη, θα έλεγα, προσέγγιση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ό,τι αφορά θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις Υπό την έννοια ότι δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε οποιαδήποτε χώρα που έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των διορθωτικών αδυναμιών της, θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να είναι πιο αποτελεσματικές, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και είμαι από την Ελλάδα, έχουμε εμπειρία, δεν κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και τώρα πληρώνουμε το τίμημα αφετέρου. Θα πρέπει να αποφύγουμε το free for all. Θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν κάποια κριτήρια ασφαλώς. Νομίζω ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λίγο πολύ σωστή. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια αξιολόγησης, λοιπόν, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε προκειμένου να μην δημιουργήσουμε πιο πολλά προβλήματα από ό,τι υπήρχαν εξ αρχής. Μπορούμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό, να το βάλουμε σε ένα έγγραφο. Δεν θα ικανοποιήσουμε τους πάντες σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι θα ικανοποιηθούν οι πιο πολλοί από τους συναδέλφους χωρίς να χάσουμε και τη γενική μα κατεύθυνση, το γενικότερο προσανατολισμό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο στα ελληνικά. Η ψηφοφορία στι 24 Ιουνίου και η Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη θα εγκρίνει την έκθεσή τη τον Ιούλιο. Στην Ολομέλεια θα περάσουμε το φθινόπωρο. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2016. Όλα τα τμήματα. Νομίζω ότι πιο σωστό να δώσουμε το λόγο πρώτα στον γενικό εσύ, γιατί τον είχα μπροστά μου. Πού πήγε. Έρχεται, έρχεται ο γενικός συζητητής. <laughs> Firstly, we would like to give you the... Να πάρετε λοιπόν πρώτα εσείς το λόγο για να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή να παρουσιάσετε τις γενικές γραμμές και μετά να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και με τον εισηγητή από την Επιτροπή Ελέγχων των Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι ήδη οι κατευθυντήριες γραμμές την 11η Μαρτίου του 2015 στην Ολομέλεια έχουν ήδη εγκριθεί. Υπεραμεινόμαστε τον της επιχειρηματικότητας, του πνεύματος επιχειρηματικότητας των, εταιριών, των επιχειρήσεων ε, και της εργασίας, ε, καθώς επίσης και την πολιτική συνοχή, αλλά βεβαίως η πολιτική συνοχή ε, συμβάλλει και αυτή στην εξωτερική αλληλεγγύη, δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή τι συμβαίνει γύρω από την Ευρώπη ε, και ε, αναφέρομαι εδώ και στην ασφάλεια και στην μετανάστευση. Κάτι σημαντικό για μας είναι ο σεβασμός των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων. Ε, συνεχώς, διαρκώς πρέπει να υπενθυμίζουμε στο Συμβούλιο ότι υπάρχει το θέμα της ευελιξίας. Δεχτήκαμε μείωση ε, για το πλαίσιο 14-20 έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ας πούμε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουμε τα χρησιμοποιητά περιθώρια τα οποία θα προσθεθούν στο συνολικό ε, ε, περιθώριο. Αυτό βεβαίως έχει σαν στόχο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα αφορούν την προστασία της εργασίας. Αναφέρομαι πούμε εδώ και στην πρωτοβουλία για την εργασία εργασία των νέων. Ε, στις 23 Ιουνίου θα, πληρώσ... θα ψηφίσουμε ε, στην Επιτροπή για την ε, για την εντολή της τριμερούς. 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη συζήτηση στην έκθεση. 22, 28, 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συζήτηση για τις τροπολογίες. 12-13 η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και τέλος τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια και μετά η Positive, positive aussi euh, και μετά στην διαλλαγή. Όσον αφορά την Επιτροπή ΕΚΟΝ, ε, η οποία έχει μοιρασμένες ε, υποχρεώσεις ε, για το Ταμείο ΕΦΣΥ, το οποίο βεβαίως θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στον ορίζοντα 2020 και στο στο μηχανισμό Connecting Europe για να μειωθεί ο αντίκτυπος αυτά τα δύο ε, προγράμματα ε, έχουμε ήδη ε, συμφωνήσει επί ενός προγράμματος το οποίο θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα και την, τις θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τώρα για ζητήματα τα οποία συνδέονται πιο στενά με τα θέματα της ΕΚΟΝ, κυρίως δε ε, όσον αφορά την ε, εποπτεία, ε, την ΕΣΜΑ ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι και για την ΕΜΠΑ και για την ΕΜΠΑ και για την ΕΣΜΑ έχουμε συγκεκριμένα κονδύλια και όσον αφορά ε, του, τις ε, πληρωμές και όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις 1,2 ε, στην μία περίπτωση για την, ε, ε και για την ΕΣΜΑ 1,7. Επίσης, μέσω των αυξήσεων αυτών δίνουμε την δυνατότητα για προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα. Ε, δεν έχουμε ε, πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο, ωστόσο είναι ένα περιθώριο το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα καθώς επίσης και για προπαρασκευαστικές δράσεις. Ε, Αυτά είναι τα κύρια σημεία. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν προγράμματα όπως το Φισκάλι, το Φίνσε, όλα αυτά αναφέρονται ε, στον προϋπολογισμό και έχουμε αύξηση σε σχέση με το 2015. Μη λησμονούμε ότι μιλάμε για το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν. Το Συμβούλιο ε, θα κάνει τη δική του ανάγνωση ε, καμιά φορά φοβόμαστε και τα χειρότερα όταν αρχίζει να διαβάζει το Συμβούλιο το προσχέδιο προϋπολογισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαφείς τουλάχιστον οι δικές μας ε, προτεραιότητες και για αυτές τις πληροφορίες ήρθα εγώ εδώ να σας δώσω, αλλά κυρίως ήρθα για να σας ακούσω και για να σημειώσω το δικό σας προβληματισμό και τις ε, δικές σας προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Πέτερ Σίμον, τον εισηγητή μας για να μας παρουσιάσει τις δικές μας ιδέες από πλευράς της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος και τον εισηγητή. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή. Θα περιοριστώ σε ένα σημείο το οποίο από πλευρά τη ΕΚΟΝ είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σε ό,τι αφορά τι τρει υπηρεσίε και ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε όλα τα θέματα, είτε στο EBA, είτε το IOPA, είτε το ESMA, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούμε ότι παρά το, τις αυξήσεις που προβλέπονται στις υπηρεσίες, ό,τι αφορά το θέμα της χρηματοδότησης για το προσωπικό, σε καμία περίπτωση δεν αρκούν τα κονδύλια. Αναφέρατε ότι έγινε αύξηση 27,7% αλλά ακούμε ότι ακόμα και οι βασικές λειτουργίες αποτελούν μια πρόκληση. Αυτό προκαλεί τρόμο. Καταρτίζουμε νομοθεσίες. Έχουμε τρεις εξαιρετικές υπηρεσίες τις οποίες ιδρύσαμε, αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση σε δύο από τις τρεις υπηρεσίες. Υπάρχει τέτοια ανάγκη στις υπηρεσίες σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την ικανότητα ανταπόκρισης στα καθήκοντά τους όπως το περιμένουμε και θέλουμε. Θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή κάτι πάει στραβά ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου έχουμε μείον φέτος σε ό,τι αφορά τη μείωση του προσωπικού. Ακούμε λοιπόν από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ευγνώμονε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα σε ό,τι αφορά ε, την, τα McDonald's, την υπόθεση McDonald's, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι πολύ απλά δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακα των συνθήκων γιατί δεν έχει το προσωπικό τα χρήματα μπορούμε να στεζόμαστε ε, σε βάθος χρόνου, σε συνδικάτα, ΜΚΟ κτλ. Να κάνουν τη δουλειά την οποία έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εμείς ε, ιδρύσαμε επιπλέον υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ακούσω και την δική σας εκτίμηση. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα εμβαθύνουμε τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει να εξαγαγούμε τα συμπεράσματά σας, ε, τα συμπεράσματά μας σε θέματα προσωπικού. Έχετε ακούσει, έχετε σχηματίσει παρόμοια εικόνα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Ποια είναι η απόψή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την εισαγωγή που θέτει κάποια ερωτηματικά. Θα τα απαντήσουμε όμως πριν το Σεπτέμβριο. Από το ΕΛΚ. Ο Παύλος Ζάλμπα. Ο Ντάριους είναι στην λίστα, αλλά δεν τον βλέπουμε στην αίθουσα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμμερίζομαι τα περισσότερα από αυτά που ακούστηκαν ε, μέχρι τώρα. Ε, ακούσαμε και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κινητικής Τράπεζας ε, πριν από λίγο να μιλάει για την ανάγκη ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να μπορέσουμε μέσω και βράχη πρόθεσμα να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος θα πρέπει να ζητήσουμε και τη στήριξη αυτών των, ε, ε, ε, αυτών των υπηρεσιών που είναι τόσο σημαντικές σε αυτή την νέα σκηνή ας πούμε των αρμοδιοτήτων. Αυτό ήθελα να σας πω και να είναι σαφές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το ECR. Λέτνε. Kiitos puheenjohtaja. Κίτος λέει ο Μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη έκθεση που αντιμετωπίζω ως χειοδής συζητήτρια στο Κοινοβούλου. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Σουίτμπορν για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει. Όπως ξέρετε, η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θέλει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πειθαρχία στον προϋπολογισμό δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να διονγκώνεται όλο και περισσότερο ο προϋπολογισμός και ότι αυτό θα οδηγήσει καλύτερα αποτελέσματα. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια στιγμή που τα Εθνικά Κοινοβούλια περιστέλουν τις ταπάρες τους, θα πρέπει και το, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το ίδιο. Πιστεύουμε ότι ο προπολογισμό του 2016 θα είναι πρέπει να το πρώτο απτό παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, έχει σημαντικό ρόλο στα σημαντικά θέματα και περιορισμένο στα μικρά πράγματα. Ο προπολογισμό θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να λύσουν τα διορθωτικά προβλήματα που τα απασχολούν με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε και στην Κομισιόν ότι το 2010 είχε τονίσει ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να <clears throat> διέπεται από την αρχή της προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή λοιπόν της προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να διατηρηθεί. Πιστεύουμε ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να σεβαστεί και την αρχή της επικουρικότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταεθνιστών δίνουν μεγάλη σημασία και εκτιμούν ιδιαίτερα την αξιολόγηση που έχει γίνει στα πλαίσια της <clears throat> χρηματοοικονομικής ε, επιθεω... Ε, εποπτείας και επισκόπησης. Πρέπει όμως τα συστήματα αυτά να είναι αποτελεσματικά ώστε να μην χρειάζεται να υπάρξει επικάλυψη των προσπαθειών που γίνονται. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει <clears throat> να έχουν προτεραιότητα ώστε να μειωθεί ο συνολικό, το συνολικό βάρος των ενεργειών και το κόστος θα πρέπει όλο να γίνεται σαφές γιατί για αυτές τις στρατηγικές επενδύσεις θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και με τους άλλους συναδέλφους στις άλλες επιτροπές και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Σάιμον και τους άλλους γεωδησίτες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα για τους φιλελεύθερους ο Νίλς Τόρβαλτς. Σας ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρε. Και μετά θα το γυρίσω στα αγγλικά. Καταρχάς, νομίζω ο, ότι από πλευρά της, υπο, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού είμαστε σε καλά χέρια. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο γενικό εισηγητή από το Χωσέ Μανουέλ που ξέρει τα μέσα και τα έξω στον προπολογισμό. Άρα από την άποψη αυτή δεν έχουμε πρόβλημα σε... κατά πάσα πιθανότητα. Ένα σχόλιο για τι υπηρεσίε και το προσωπικό. Νόμιζα ότι την ίδια συζήτηση την κάναμε και πριν από ένα χρόνο. Και αν δεν κάνω λάθος, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό τους και για το 2015. Αλλά αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Και αυτό γιατί χρειάζονται προσωπικό, καλό προσωπικό και θα ήταν καλό και θετικό να τους κάνουμε μία αξιολόγηση. Πόσα άτομα κατάφεραν να πάρουν επιπλέον για να κατανοήσουμε με καλύτερο τρόπο γιατί ποσά μιλάμε, τι ποσά χρειάζονται τα επόμενα χρόνια. Ένα σύντομο σχόλιο τώρα από δικής μου πλευράς ένα κλασικό πολιτικό πρόβλημα. Κοιτώντας όλες τις προτεραιότητες. Είμαστε εξαιρετικοί στο να θέτουμε προτεραιότητες. Όταν οι προτεραιότητες διωγγώνουν τον προϋπολογισμό. Όταν όμως πρόκειται για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού και τις περικοπές ε, κάποιων προγραμμάτων, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, όσο όταν βάζουμε κάτι στη λίστα, κάτι που θέλουμε, θα έπρεπε παράλληλα να βρούμε και κάπου να κάνουμε περικοπές. Ιδάλλως, θα κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση στην οποία έχουν βρεθεί κάποια κρατημέλη, σε έναν προϋπολογισμό δηλαδή, το οποίο δεν θα είναι συσκελισμένος. Αυτό δεν το θέλουμε. Αυτά από δική μου πλευρά και σα ευχαριστώ πολύ στα γερμανικά. Σα ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο, και τώρα από του πράσινου να δώσω το λόγο στον Σφεν Κίγκολτ. Είναι η σειρά μου. Ωραία. Θα ήθελα να πω λοιπόν το εξή. Κανονικά η αριστερά δεν προηγείται. Α, συγγνώμη. Ε, στον κατάλογό μου σε πρώτο. Εγώ το κατάλογο ακολουθώ. Αν έτσι λέει ο κατάλογο ε, και ο κατάλογο είναι από τη γραμματεία, θα προσευχηθούμε και θα πούμε ότι είναι σωστό. Μάλιστα, πολύ ωραία, δεν θα φέρω αντίρρηση. Συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ για το θέμα αυτό. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια συγκεκριμένα σημεία. Όντω γνωρίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες αυτές υπάρχει αντίφαση ότι τους δίνουμε όλο και πιο πολλές ε, αρμοδιότητες και ε, σε πολύ περιορισμένο βαθμό προσαρμόζουμε τον προϋπολογισμό και η επιστολή της ΕΙΟΠ αποτελεί λόγο ανησυχίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο. Η κοινή επιτροπή των ε, τριών υπηρεσιών μας, να μας παρουσιάσει την κοινή θέση, την κοινή της άποψη για το θέμα αυτό. Ίσως θα μπορούσε να το ζητήσουμε αυτό από πλευρά της ομάδας μας. Κατά δεύτερον, εκ παραλίλου, συζητάμε τον προπολογισμό και η στιγμή είναι σωστή για να θέσουμε κάποια προβλήματα, κάποιε προβληματικές εξελίξεις. Δεν έχω υπόψη μου την ΕΙΟΠΑ γιατί δεν έχουν πολλέ νομοθετικέ αρμοδιότητε ακόμα. Αλλά προσφάτω είδαμε στην ΕΣΜΑ ότι το Κοινοβούλιο, η ομάδα του Κοινοβουλίου τη οποία ηγείται ο πρόεδρο Φέρμπερ, δεν έτυχε ευνοϊκής αντιμετώπισης και όλο και πιο συχνά παρατηρείται ότι όταν οι επιτηρητές συμφωνούν επί κάποια θέση στο εποπτικό σώμα, εμείς εκ των υστέρων ερχόμαστε και δεν υπάρχει διάθεση να ληφθεί υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά συζητήσεις που έγιναν με την EBA. Δεν ήταν πολύ απλό να το θέσω με κόμψο τρόπο να θέσουμε τις ανησυχίες μας. Ίσως λοιπόν αυτή τη χρονική στιγμή του προϋπολογισμού θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τις υπηρεσίες αυτές πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει αποτελεσματικά στην νομοθετική διαδικασία και σε μετέπειτα χρονική στιγμή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την δυνατότητα α, τοποθέτησης κάποιων τμήματων του προπολογισμού στο αποθεματικό. Κατά δεύτερον, με τη Eurostat, όταν ήμουν εισηγητής για το θέμα αυτό, τους έθεσα θέματα ποιότητας στα στατιστικά τους στοιχεία. Λάβαμε κνέου μια ενημέρωση για τους στόχους για το 2020, τη βασική στρατηγική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε κάποια αριθματικά στοιχεία για το 2013 για τους έξι βασικούς δείκτες, τα οποία δεν διατίθενται ακόμα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί δεν είναι σε θέση η Eurostat να μας δώσει στατιστικά δεδομένα που θα μας βοηθήσουν πραγματικά να καθοδηγήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους δείκτες αυτούς, για παράδειγμα. Αυτό είναι η βασικό τους καθήκον. Ε, διάφοροι δείκτες, λοιπόν, δεν διατίθενται. Νομίζω ότι τα θέματα ποιότητας που αντιμετωπίζει η Γιουρούστα θα πρέπει να τεθούν. Μία ερώτηση τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του ΕΦΡΑΚ και του ISB. Προβλέπετε σημαντικές αυξήσεις. Μου προκαλέσε μία κάποια έκπληξη αυτό. Γιατί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ISB, ξέρουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκλέγεται δημοκρατικά. Και οι Ευρωπαίοι στο Συμβούλιο αυτό δεν εκλέγονται δημοκρατικά. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις που ε, θέτουν πρότυπα σε θέματα ε, λογιστικής. Γιατί λοιπόν αυτή η σημαντική αύξηση των κονδυλίων και τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρχει πιο δημοκρατική ε, εκπροσώπηση στο όργανο αυτό. Και τέλο, συμφωνώ απόλυτα με τον Πέτερ Σίμων σε ό,τι αφορά την ανάγκη να υπάρχουν μεγαλύτερε ικανότητε σε θέματα φορολογικά. Έχουμε το πρόγραμμα φυσκάλη, το οποίο αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εφοριακών αρχών. Ξέρουμε ότι γίνονται όλο και πιο πολύ διασυνοριακοί έλεγχοι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των φορολογικών ζητημάτων και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνώ απόλυτα δε ότι δεν θα πρέπει να, να επαφιόμαστε στα συνδικάτα να ερευνούν τα φορολογικά προβλήματα της εταιρείας McDonald's. Αυτό καταδεικνύει πασίφανο ότι λείπουν κονδύλια, λείπουν, λείπει χρηματοδότηση. Αν λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι προ την κατεύθυνση αυτή, εμεί έχουμε καταθέσει ένα πολιτικό έργο, ίσω θα μπορούσαμε να εντάξουμε κάποια στοιχεία για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Και θα ήθελα να κατανοήσω και πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αύξηση χρηματοδοτήσεων προ ένα σύστημα το οποίο δεν έχει δημοκρατική εκπροσώπηση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να σας δώσω προτεραιότητα εναντί άλλων πολιτικών ομάδων και να σας δώσω και άλλες έδρες στην ομάδα των Πρασίνων. Όχι, όχι, αυτό δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου, λέει ο κύριος Φέρμπερ. Συγγνώμη θα δώσω το λόγο στον Μιγγέλ Ούρβαν Κρέσπο για την ΚΟΕ. Δεν έχω πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μας ομάδα δεν ε, συμμερίζεται αυτή την θετική αξιολόγηση που κάνετε στο πρόγραμμα Juncker γιατί ε, αυτού του είδους η αντιμετώπιση των κεφαλαίων για την εμπόσχα της κρίσης ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θέλουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή τι είδους δραστηριότητες θα συμπεριληφθούν, με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν κτλ. Όσον αφορά τις επενδύσεις, φαίνεται ότι ε, θα υπάρχει μεγάλη επικέντρωση των επενδύσεων που, ε, στις οποίες θα λάβουν χρήματα ε, μεγάλες πολυεθνικές. Στα πλαίσια του τελευταίου προγράμματος COSME εμείς θα θέλαμε να δούμε τέτοιου είδους επενδύσεις, κυρίως με τρόπο ώστε η επιχειρηματικότητα η οποία θα ε, ε, τονωθεί, να είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινωνικά αλληλέγγυα ε, οικονομία. Ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η κοινωνική ισορροτιμία ε, και η κοινωνική ε, και η ισορροπία ε, μεταξύ των πολιτών. Δεν εμείς θα θέλαμε επίσης να δούμε κάποιες εμπροστοβαρείς πληρωμές σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την νεανική ανεργία έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτήν την νεολαία ε, η οποία βρήκε κλειστές πόρτες μέχρι τώρα. Ε, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ε, χτίζουμε αυτήν την Ευρώπη φρούριο, ε, πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις νέες μορφές και τα νέα κύματα μεταναστών που δεν είναι μονάχα οικονομική μετανάστευση αλλά είναι μετανάστες που έχουν ξεκινήσει από χώρες που αντιμετωπίζουν πολέμους κτλ. Εμείς θέλουμε να ενισχυθούν οι δημοκρατικές και κοινωνικές κοινωνικές αρχές οι οποίες θα αφορούν όλο τον κόσμο και πολιτικές οι οποίες ε, θα είναι κοινωνικά δίκαιες και θα αφορούν ολόκληρο τον κόσμο στα πλαίσια των, ε, της ε, χρήσης των, του κοινωνικού ταμείου. Επίσης η χρήση πόρων για την γεωργία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους στόχους για την πράσινη ανάπτυξη και για τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε κατά πόσον ταυτίζονται με τους στόχους αυτούς ε, αυτά τα σχόλια, τα οποία, ε, συγγνώμη, αυτά τα προγράμματα τα οποία αφορούν τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ταυτίζεται η αντιμετώπιση που θα έχουμε των οικονομικών προγραμμάτων κυρίως για χώρες οι οποίες είναι πλούσιες και οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ένα σύστημα επιστροφών και εκπτώσεων που τους οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερα έσοδα. Εμείς επίσης δεν θέλουμε να δοθούν χρήματα σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει το φορολογικό ε, dumping ε, ή ε, την κίνηση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Ε, θα θέλαμε επίσης να ενισχυθεί ε, η σωστή αντιμετώπιση των εργασιακών πολιτικών από πλευρά της Ευρώπης για τους εργαζόμενους της Ευρώπης. Ε, εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τους ανθρώπινους πόρους και την, ε, την επαγγελματικότητά τους. Θέλουμε ε, να έχουμε καλύτερες θέσεις εργασίας και όχι περικοπές και μειώσεις των θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το EFTD. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Βλέπω ότι εξετάζεται να μειώσετε το κόστος στους τομείς. Στους τομείς αυτούς όπου απαιτούνται εξοικονομήσεις και εγώ θα ήθελα περιμένω να ακούσω και την άποψη του κυρίου Σάιμον την θέση του γιατί αυτός θεωρεί ότι για τις τρεις αυτές ε, υπηρεσίες, την Υπηρεσία Αγορών και Αξιογράφων και την ε, Τραπεζική Αρχή και την Αρχή για τα Ασφαλιστικά, πρέπει εκεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση κατά την άποψή μου. Βέβαια, όταν σφίγγουν το ζωνάρι τους οι πληθυσμοί της Ευρώπης σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει να έχουμε μια πιο μεγαλύτερη υπευθυνότητα για το κόστος προς τους φορολογούμενους που πρέπει να ελέγξουν όλα αυτά τα θέματα. Εμείς θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την πορεία χρηματοδότησης και συμφωνούμε με τον κύριο Τίμερμαντς και τον κύριο Γιούγκερ ότι πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση των προγραμμάτων αυτού του είδους και φυσικά όλοι οι δημόσιοι φορείς μεταξύ των οποίων και αυτοί οι τρεις ε, φορείς θέλουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους και να λένε ότι θέλουν περισσότερους ανθρώπους. Αλλά εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει η αρχή της επικορικότητας εδώ. Υπάρχουν κάποιοι φορείς, παραγωγός στη δική μου χώρα υπάρχουν πολύ σημαντικοί και ισχυροί ρυθμιστικοί φορείς που μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη. Θα πρέπει να σκεφτούμε να κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες ώστε ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερος. Αυτά είναι τα αρχικά μας σχόλια λοιπόν κύριε Πρόεδρε και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη σύνολη διαδικασία. Ευχαριστώ. Λέω ο πρόεδρο. Έχουμε ακούσει όλε τι πολιτικέ ομάδε Και η κυρία Μάλετιτ έχει ζητήσει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Να αναφέρω <clears throat> ότι εμάς μας ενδιαφέρει για τους τρεις αυτούς φορείς να αντιμετωπιστεί σωστά ο προπολογισμό τους, αλλά όχι μόνο για αυτούς τους τρεις προαναφερθέντες φορείς. Μας ενδιαφέρει σωστή οικονομική διακυβέρνηση, και όλα τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την καλή οικονομική διακυβέρνηση και οι προϋποθέσεις είναι η σωστή οικονομική διαχείριση, οι έγκαιρες πληρωμές και στην υγεία χρηματοδοτική διαχείριση. Τονίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλες οι συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με το θέμα αυτό, είτε πρόκειται για λογιστική, για στατιστική, για φορολογία, μιλήσατε για το Φισκάλης και το Ηρακλή και θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων θα μπορέσει να προχωρήσει και κατά πόσο θα έχει αυτό αντίκρισμα στον προϋπολογισμό σε σχέση με τις έγκυρες πληρωμές. Νομίζω ότι ως Επιτροπή ΕΚΟΝ θα πρέπει να σκεφτούμε τα προγράμματα <clears throat> τα οποία αναμένουν ακόμα πληρωμές, προγράμματα στον τομέα της συνοχής, γιατί αυτές οι καθυστερήσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο, δημιουργούν προβλήματα ρευστότητα στα κράτη-μέλη. Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα μόνο της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων, αλλά και της δικής μας Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο εισηγητής δεν θέλει το λόγο. Και ο, ξαναδίνω το λόγο στον Ζωζέ Μανουεό, αν θέλει να πει κάτι. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο. Να μην λησβονούμε ότι η Κομισιόν ε, παρουσίασε το προσχέδιο προϋπολογισμού και τώρα θα μελετηθεί ο προϋπολογισμός αυτός. Βεβαίως ε, είναι ένας μικρός προϋπολογισμός, 1% ε, του ΕΕΠ, 55 δις ευρώ περίπου. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος παρά τους προβληματισμούς, παρά την αύξηση των μελών μας, το τώρα 28, παρά την δημιουργία νέων υπηρεσιών, παρά το, τις νέες αρμοδιότητες που έχουμε, παρόλα αυτά λοιπόν παραμένει στο 1% του ΑΕΠ και βεβαίως αυτό μας ε, οθεί στο να έχουμε ε, ιδιαίτερα υψηλή αποτελεσματικότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε τους συμβιβασμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις, θα πρέπει να σεβαστούμε τον πολιετή προγραμματισμό, αλλά ωστόσο ταυτόχρονα θα πρέπει οι διάφορες υπηρεσίες να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα τους επιτρέψει να κάνουν την εργασία που πρέπει και οφείλουν ε, γιατί έχουν δεσμευτεί να ε, κάνουν. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε βεβαίως, ε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την Επιτροπή ΕΚΟΝ με στόχο τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς ε, τους οποίους υφιστάμεθα. Ε, μιλήσαμε εδώ για τρεις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά ξέρουμε ότι για το πρόγραμμα φυσκάλης και, τα, και άλλα τα άλλα προγράμματα είναι προγράμματα στα οποία οι δεσμεύσεις εκτέλεσης των διαφόρων υπηρεσιών είναι της τάξης του 100% όσον αφορά τις πληρωμές. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Θα έχουμε βεβαίως μετά και την εντολή για τον τριμερή διάλογο, για τους τριμερείς διαλόγους μάλλον. Θα δούμε και τις τροπολογίες. Θα δουλέψουμε όλοι στενά έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες ε, των ε, ε, πολιτών αλλά και τις προσδοκίες εδώ της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Επόμενη ανταλλαγή απόψεων από τις εκθέσεως αυτής, 15-16 Ιουλίου. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 13 Ιουλίου το μεσημέρι. Ίσα ίσα πριν φύγετε για διακοπές συζήτηση επί των, προϋπολογισμών, ε, επί των <laughs> τροπολογιών συγγνώμη, 3 ε, Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να υπολογίσουμε το χρόνο έτσι ώστε οι τροπολογίες μας να φτάσουν έγκαιρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεύτερη, ε, η δεύτερη σύνοδος του Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου για την Ολομέλεια. Η Κομισιόν δεν είχε ζητήσει το λόγο, δεν είχα δει κάποιον... Για τα πρακτικά να πω ότι η Κομισιόν δεν παρακολούθησε τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Ε, πράγμα ιδιαίτερος ασυνήθιστο πρέπει να πω. Θα καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Άψογα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 το πρωί.